γι' αυτό. Allora, riprendiamo formalmente la nostra seduta. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Να Έχουμε στην ημερήσια διάταξη. Την κυρία Μακλέιρ. την καθηγήτρια Ζάκλιν Μακλέιρ, η οποία επρόκειτο να παρευρεθεί ως Executive Director του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Είχε παρευρεθεί στην Επιτροπή μας και πριν από δύο χρόνια. Και θα μας παρουσιάσει σήμερα εκ νέου την ε, θέση της αναφορικά με τις ε, επιδόσεις της πολιτικής ε, περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις ε, μεταφορές. Με την έκθεση λοιπόν αυτή θα λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για τα θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα και επανειλημμένα. για τους στόχους που μας απασχολούν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, τους οποίους επιδιώκουμε. Για τη διαμόρφωση δηλαδή της κινητικότητας με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Και σε αυτό το σημείο συμπεριλαμβάνεται και η βιώσιμη αλλά και η ασφαλής κινητικότητα. Αυτή είναι η στόχη μας στην Επιτροπή Μεταφορών. το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να κοιτάξουμε ένα τέτοιο κείμενο το οποίο είναι ενημερωμένο είναι πολύ χρήσιμο για μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να συζητήσουμε την παρουσίαση αυτή πρωτού περάσουμε στη συζήτηση της έκθεσης για τα slots. Άρα, χωρίς ε, περαιτέρω τη στέρηση θα δώσω το λόγο στη Ζάκλιν Μακλέιτ για να παρουσιάσει την έκθεση της, την οποία σίγουρα θα, θα παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή. Να σας παρακαλέσω να, να αναφέρετε ό,τι θέλετε για τα θέματα αυτά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μετά από δύο χρόνια. Ελπίζω να είναι εξίσου έντονη η συζήτηση όσο και πριν από δύο χρόνια, γιατί ήταν πολύ χρήσιμο τότε να ακούσω και τις δικές σας απόψεις, αλλά και τι απόψει τη Επιτροπή περιβάλλοντο. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσει να ακολουθήσει μια ζωηρή συζήτηση. Προφανώς, πυρήνα ε, τη εργασία σα είναι το ότι οι συζητήσει για την οικονομική κρίση αφορούν τόσο πολύ το χρηματοπιστωτικό τομέα, αλλά και τον τομέα των βιομηχανίας, η... της αυτοκινητοβιομηχανίας και το σύστημα των μεταφορών. Αλλά θα ήθελα να τονίσω με την έκθεσή μου αυτή ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομικής αυτής δραστηριότητα και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον αλλά και σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί βασικά ανησυχία το θέμα του άνθρακα, το οποίο αν θέλετε συζητιέται πάρα πολύ και όπως ξέρετε και στην Κοπενχάγη θα συζητηθούν τέτοια θέματα, αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε και πάλι το αδιαφυσβήτητο ζήτημα, το ότι η βασική πηγή του άνθρακα είναι οι μεταφορές. Συνολικά οι μεταφορές βασίζονται σε ένα μη βιώσιμο πλέον μέλλον σε ό,τι αφορά και την οικονομία μας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υπάρχει δυσανάλογος αντίκτυπος ε, των μεταφορών και σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του περιβάλλοντος και σε ό,τι αφορά την ηχορύπανση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην έκθεση είναι να εντοπίσουμε κάποια από τα, κάποιες από τις ενδείξεις, αν θέλετε, τις πρώιμες, κάποιες από τις μακροπρόθεσμες τάσεις για να αμβλύνουμε κάπως τον αντίκτυπο στην αγορά και να κοιτάξουμε και ποιες είναι, ποια είναι τα μακροπρόθεσμα μηνύματα. Το 2000 είχαμε την ετήσια έκθεση για το περιβάλλον και θεωρώ ότι αυτό μας φέρνει, αν θέλετε, σε επαφή με τις άλλες, το με τις άλλες πολιτικές. Να σας πω ποια είναι τα βασικά μηνύματα, λοιπόν. Καταρχάς, οι ελεύθερες μεταφορές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ναι, ναι, θα επανέλθω στο θέμα αυτό που αναφέρθηκε εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Αυτό θα μπορούσε ασφαλώς να, αποτελεί, να αποτελέσει τη λύση. Ίσως λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό πρωτού επιτρέψουμε στα φορτηγά να επανέλθουν στους οδούς. Η ελεύθερη λοιπόν μεταφορά αυξάνεται κυρίως για τις αερομεταφορές και για τις οδικές μεταφορές. Ο συνολικός όγκος αυξήθηκε κατά 35% πρέπει να σας πω από το 1996 μέχρι το 2006. Φυσικά δεν έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία για τα τελευταία δύο έτη και είμαι σίγουρη ότι πολλές συζητήσεις θα γίνουν για το θέμα αυτό. Η ε, χώρες, αν είχαν ε, οι χώρες καλύτερη συνεργασία με τη Γυροστό, θα είχαμε καλύτερα στοιχεία και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό, αν θέλετε, την υποχρέωση υποβολής αναφορών. Γιατί φυσικά τα κράτη-μέλη όντως θα πρέπει να εργάζονται με πιο ε, υπεύθυνο τρόπο στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις συνδροδρομικές μεταφορές και τις πρωτές μεταφορές μειώθηκαν την ίδια περίοδο. Αυτό λοιπόν υποδεικνύει ότι δεν προωθούνται τόσο πολύ οι συνδρομικές και πλεκτές μεταφορές. Θα υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα δεδομένα η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία έχουν αλλάξει τη μεθοδολογία τους. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και η Eurostat δεν μπόρεσε λοιπόν να δώσει ένα διαφορετικό παράγοντα εναρμονισμένο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το ίδιο. Αλλά υπάρχουν συζητήσεις για την ε, υποβολή αναφορών. Βλέπουμε ότι επίσης αυξάνεται η ιδιοκτησία των αυτοκινήτων Στους, στην Ευρώπη των 27. 22% ήταν η αύξηση. Η χρήση των αυτοκινήτων κατά 18% και τα χιλιόμετρα που ταξιδεύουν οι άνθρωποι, οι επιβάτες, αυξήθηκε κατά... Επίσης κατά μεγάλο ποσοστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια γενικότερη τάση και φυσικά βλέπουμε ότι ο κόσμος μπορεί να απορροφήσει ε, μεγάλο υψηλό κόστος και τώρα αναρωτιόμαστε με την παγκόσμια κρίση αν θα υπάρξει αντίκτυπος και σε διαφορά αφορά τις μεταφορές των δημοτών. Ε, σε ό,τι αφορά τα αέρια του, του θερμοκηπίου. Ίδια τα πράγματα πολύ φοβούμε, αλλά έχουμε το στόχο του 20-20-20 τώρα και θα πρέπει πλέον οι εκπομπές που προέρχονται από του, τις μεταφορές έχουν αυξηθεί κατά 27% σε σχέση με τη βάση που λαμβάνει το πρωτόκολλο του Κιώτο και αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την διεθνή αεροπλοεία και ναυτιλία. Αν τις συμπεριλαμβάναμε και αυτές θα ήταν 36% το ποσοστό αυτό. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε. Να περάσω στην ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας τώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κατεπήγον θέμα που μας απασχολεί. Η ρήπανση της ατμόσφαιρας είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά ε, τα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Για να σας δώσω μια τάξη κλίμακας, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε το πακέτο για το, την ενέργεια να αποδώσει, θα μιλούσαμε για μείωση περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανά έτος σε ό,τι αφορά το κόστος δηλαδή για να ανταποκριθούμε στην νομοθεσία για τις εκπομπές. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρήπανσης της ατμόσφαιρας και τα αριθμητικά στοιχεία αυτά είναι ε, πιστοποιημένα και έχουν ελεγχθεί και από τα κράτη-μέλη. Γιατί και η χορύπανση είναι θέμα. Μιλάμε δηλαδή για 67 εκατομμύρια ανθρώπους που, 25% του πληθυσμού που εκτίθενται σε πάνω από 65 δεσιμπέλ. Δηλαδή μιλάμε για υψηλά ποσοστά. Για παράδειγμα, σαν να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, σαν να υπάρχει κίνηση αυτοκινήτων σε μικρή απόσταση κοντά σε κάθε άτομο. Μιλάμε για σημαντικούς ε, παράγοντες που βλάπτουν την υγεία. Άρα, είτε μας αρέσει είτε όχι, η υγεία βλάπτεται και από την ηχορύπανση και από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και πραγματικά είναι τεράστιο το κόστος ε, που συνεπάγονται για το υγειονομικό σύστημα. Είτε μας αρέσει λοιπόν είτε ή όχι, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά, να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Κοιτώντας λοιπόν και άκουσα και τι έγινε χθες για τη συζήτηση με την ε, Ευρωβινιέτα, υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα πράγματα τα οποία θα πρέπει να παρατρύνουμε θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τον αντικτύπο των μεταφορών για όλους τους τρόπους μεταφορών, αλλά κυρίως για τις οδικές μεταφορές. Θα πρέπει να περιορίσουμε τον περιβαλλοντικό αντικτύπο και θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο που μεταφέρεται στην Ευρώπη ε, τα εμπορεύματα. Όλα, όλοι οι τρόποι μεταφορών θα πρέπει να συμπεριληφθούν και σίγουρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πώς θα ενεργήσουμε σε ό,τι αφορά τις πόλεις για την ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα, και για το πώς γίνεται η αστική μετακίνηση, οι αστικές μεταφορές. Σε ό,τι αφορά και για παράδειγμα την αποδοτικότητα των οχημάτων. Να κοιτάξουμε τώρα την αποδοτικότητα των καυσίμων και των οχημάτων. Τα βιοκαύσιμα ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία 12, 12 μήνες. Στο κλιματικό πακέτο, σε ό,τι αφορά δηλαδή τους ε, κανόνες που πρέπει να οριστούν για την βιώσιμη ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυξάνεται η χρήση του ντίζελ και τα δηληστήρια, αν θέλετε, δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές, το οποίο θα μπορούσε να έχει συνέπεια στις θαλάσσιες ε, μεταφορές. Τα βιοκαύσιμα όμως δεν αποτελούν και αυτά λύση, γιατί αυξάνεται η τιμή τους Άρα ούτε αυτά θα μείνουν πίσω σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών, σε ό,τι αφορά την ε, αποδοτικότητα των οχημάτων τώρα. Δεν υπάρχει μεγάλη πρόεδρος, υπάρχει ο κανονισμός για τα 130 γραμμάρια ανά χιλιόμετρα, αλλά από ό,τι ξέρετε το θέμα είναι η θέρμανση των καθισμάτων, τα air conditioning κτλ. Άρα θα πρέπει να επηρεάσουμε τις επιλογές των καταναλωτών, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την οικοσήμανση και ούτω καθεξή. Και δεν έχει σημειωθεί πρόοδο, θεωρώ, τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, κοιτώντα και του κανόνε για το καμποτάζ και πώς θα προχωρήσει αυτό στο μέλλον, θα ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια στιγμή που θα πρέπει να περάσουμε από την προσέγγιση μας την επιθετική στο πώς θα περιλάβουμε τις μεταφορές στο πακέτο της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Κάτι θα πρέπει να γίνει και με τη φορολογία. Και κάτι θα πρέπει να γίνει για να αντισταθμιστεί το κόστος ε, των μεταφορών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Δεν θα ήθελα να πλατιάσω κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό προτιμώ να σταματήσω τώρα και να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το σύνολο της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Μαγκλέιτ. Πραγματικά οι προτάσεις σας θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για μας. Εγώ δεν έχω προσωπικά σχόλια, δεν θέλω τουλάχιστον να κάνω προσωπικά σχόλια αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων των μελών της Επιτροπής Μεταφορών στο γεγονός ότι το περιεχόμενο της έκθεσης, ε, κάποια στοιχεία θα μας αρέσουν και κάποια ίσως όχι, ολόκληρη η έκθεση όμως μας βοηθά και ελπίζω να βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση. Το ίδιο και οι ενδιαφερόμενοι. Θα πρέπει να αντιληφθούμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών χωρίς ε, να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα των μεταφορών. Είναι αδύνατο να επιλύσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποκλείοντας τις μεταφορές από τη λύση. Και όσες φορές προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ευαισθητοποίηση για τη σημασία των μεταφορών στον προβληματισμό του περιβάλλοντος, αντιληφθήκαμε πόσο δύσκολο είναι. Είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε δυσκολίες με την παράταση για παράδειγμα των επεμβάσεων στις υποδομές από το πακέτο κινήτρων για την ζήτηση στις υποδομές των μεταφορών. Η Κομισιόν δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας. Παρ' όλα αυτά, είναι προφανές ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα αποφέρουν καρπούς. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από τη συμπερίληψη των μεταφορών στην προσπάθεια αντιμετώπιση των ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων. Και θα πρέπει να βρούμε κάποια κοινά σημεία μέσω των στόχων, των αναγνωρισμένων στόχων της κινητικότητας, για παράδειγμα. Έχουμε κοινά στοιχεία. Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί όλοι θέλουμε ασφαλείς, αποτελεσματικές και βιώσιμες μεταφορές. Είναι πολύ χρήσιμη λοιπόν ως προς αυτό η ετήσια έκθεση, παρόλο που ίσως ορισμένα σημεία της θα μας δυσαρεστήσουν. Θα έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων, πρώτα ο κύριος Γιωζεμπόφσκι. Αξιότιμη κυρία καθηγήτρια, θα ήθελα φυσικά να διαβάσω την έκθεσή σας. Θα ήθελα όμως να κάνω και κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε. Πάντα με δυσαρεστεί το γεγονός όταν όλοι τα βάζουν με τις μεταφορές, γιατί κανείς δεν βγαίνει να μιλήσει για το πώς η ρήπανση προκαλούν τα νοικοκυριά, για παράδειγμα. Ένα μεγάλο τμήμα, ένα τρίτον της παγκόσμιας ρήπανση τουλάχιστον, προέρχεται από τα ιδιωτικά νοικοκυριά και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αχ, σταματήστε πια, σταματήστε, ρωτήστε τι συμβαίνει πραγματικά. Θα μιλήσεις μετά, μετά να μιλήσεις εσύ, όταν ήρθε η σειρά σου. Θα έρθει η σειρά σου μετά. Είναι τρομερό πάντα δηλαδή πόσο τα βάζουμε με τις μεταφορές πάντα. Μπορούμε να συζητήσουμε και τα συστήματα εμπορίας ε, ρήπων της βιομηχανίας αλλά και τα νοικοκυριά που οφείλεται και μεγάλο ποσοστό της ρήπανσης. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι το στο τομεακό επίπεδο κάναμε κάποια πράγματα στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι το σύστημα εμπορία ρήπων, το οποίο αποφασίσαμε μαζί με το Συμβούλιο για το θέμα των ε, εναέριων μεταφορών, ήταν πραγματικά υποδειγματικό. Και προσπαθούν τώρα να πείσουν τους Αμερικανούς να κάνουν ε, το ίδιο. Δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο, μπορεί ο Ομπάμα να δείξει κάποια προθυμία, αλλά εγώ τηρώ διστακτική και επιφυλακτική στάση. Άρα θα πρέπει να επενέσουμε το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις ενέργειες μεταφορές το Συμβούλιο έλαβε σωστή απόφαση. Νομίζω ότι με το ETS έχουμε ένα καλό εργαλείο για την αγορά. Το βασικό μου πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι αποφασισμένη. Ε, ήμουν ε, υπεύθυνο για μια έκθεση για την πιο πράσινη διαμόρφωση των μεταφορών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα και το Κοινοβούλιο κατάφερε να εντοπίσει τα πιο πολλά ε, στοιχεία, αλλά είναι πάρα πολύ διστακτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Τέλος Κυκλοφορίας, την Ευρωβινιέτα. Θα εισάγουμε αυτό το μέτρο Είτε θα δεχτούμε τη λογική της παροχής ε, κινήτρου μέσω τιμών για την ε, ανανέωση των οχημάτων, είτε όχι. Ας το κάνουμε τότε και στους άλλους ε, τομείς μεταφορών που θα έπρεπε και αυτοί να τους εξετάσουμε. Η Κομισιόν σε αυτούς τους τομείς δεν κάνει τίποτα. Για παράδειγμα, ένα σύστημα ETS για την αυτιλία δεν υπάρχει καθόλου τίποτα τέτοιο. Γιατί δηλαδή μιλάμε για την ε, εσωτερικοποίηση του εξωτερικού κόστους για τα φορτηγά και όχι για τα άλλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις προτάσεις της δεν ακολουθεί ένα συστηματικό και δίκαιο τρόπο και δεν ε, ανταποκρίνεται σωστά στην κατάσταση. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το εξή. Κάθε έκθεση, όπως είπατε, αποτελεί μια χρονικά περιορισμένη έκθεση. Από την άποψη λοιπόν αυτή, τα συμπεράσματα για τη σημερινή κατάσταση αυτή είναι λίγο παροχημένα, γιατί στην εναέρη κυκλοφορία έχουμε μείωση του 30% για τους επιβάτες 5-10% μείωση. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εκθέσουμε και να δούμε αν οι μειώσει αυτές έχουν νόημα αν είναι σκόπιμες, γιατί μπορούμε να χαρούμε που δεν υπάρχουν για παράδειγμα σε αέριες μεταφορές εμπορευμάτων, αλλά αυτό από την άλλη πλευρά τι σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπορεύματα, υπάρχει ανεργία στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Ταϊβάν, δεν ξέρω πού. Αυτό που προσπαθώ λοιπόν να σας εξηγήσω είναι το εξής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι η κατάσταση στην πραγματικότητα. και να δούμε τι θα ήταν οικονομικά σκόπιμο. Για παράδειγμα το σύστημα ETS, για τις ενέργειες μεταφορές. Είναι κάτι που μπορεί να αποδεχτεί ο κλάδος. Για το τέλος συμφόρηση στην Ευρωβινιέτα. Είναι υπερβολική επιβάρυνση του τομέα, γιατί θεωρώ ότι στη φάση αυτή έχουμε προβλήματα να κρατήσουμε τη θέση μα μας καν. Άρα, τελικό συμπέρασμα, θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη, όλα αυτά τα στοιχεία για το περιβάλλον, αλλά θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να καταρτίζει εξαιρετικέ εκθέσεις και να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για τις μεταφορές και για το περιβάλλον. Ο κύριος Στόκμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια για την έκθεσή της. Διαπιστώνουμε ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε πραγματικά, πρέπει όντως να δράσουμε προκειμένου και οι μεταφορές να συνδράμουν στη μείωση των εκπομπών και της επιβάρυνσης της περιβαλλοντικής, προκειμένου να καταστούν πιο βιώσιμοι οι μεταφορές. Θα πρέπει λοιπόν καταρχάς να πούμε ότι οι μεταφορές που είναι το μέσο για την ε, λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Το χρειαζόμαστε λοιπόν τις μεταφορές αυτές για την ενιαία αγορά. και θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποιους όρους. Καταρχάς την αποδέσμευση την οποία αναφέρατε, η οποία φυσικά θα πρέπει να υπάρξει, αλλά αυτό εξαρτάται και από την παραγωγή και από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό λοιπόν που καταλαβαίνουμε με την αποδέσμευση είναι το αντίθετο. Ο δεύτερος μύθος είναι η μετεγκατάσταση της μεταφορά, των μεταφορών. Το θέλουμε αυτό, αλλά βλέπουμε στην πράξη ότι δεν συμβαίνει. Εφόσον όμως καταβάλουμε τόσο μεγάλη προσπάθεια, δεν σημαίνει ότι δεν το θέλουμε αυτό. Το είδαμε και στο Μαρκο Πόλο, ότι πετύχαμε, δεν λειτουργούν τόσο απλά τα πράγματα. Και κατά τρίτον, η πρόληψη της κυκλοφορίας και αυτό αποτελεί ευσεβή πόθο, τον οποίο όμως πραγματικά, ρεαλιστικά δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ωστόσο κάτι πρέπει να κάνουμε, όπως είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι καταρχάς θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε αυτό το μέσο των μεταφορών και έχουμε τις τρεις γνωστές στρατηγικές και τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις στρατηγικές, την απελευθέρωση την οποία σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά το καποτάζ. Αν δεν υπήρχε ο κοινωνικός ε, προβληματισμός θα το καταργούσαμε δεν θα είχαμε κενά φορτία και θα ήταν απλά τα πράγματα, αλλά έχουμε τα εμπόδιο αυτό. Κατά δεύτερον, η στρατηγική εναρμόνισης που θα μας απασχολεί στα επόμενα 15 χρόνια τουλάχιστον, προκειμένου και ο σιδηρόδρομος, για παράδειγμα, να κινείται χωρίς σύνορα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές εμπορευμάτων. Γιατί στα εμπορεύματα έχουμε τις μεγάλες ε, αυξήσεις και σε ό,τι αφορά τη στρατηγική ενοποίησης έχουμε ακόμα μεγάλες διαφορές. Όλα αυτά ακούγονται θεωρητικά καλά, αλλά στην πράξη δεν λειτουργούν. Και καταλάβαμε πλέον ότι θα πρέπει να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, να, κοιτάξουμε από τα, να ξεκινήσουμε από τα ευφύη συστήματα και όχι από άλλες διαπαφές οι οποίες κοστίζουν πολύ και δεν λειτουργούν ενδεχομένω τόσο καλά. Άρα θεωρώ ότι στις μονομένες στρατηγικές υπάρχει δυναμικό Σημαντικό είναι να συνεχίσουμε με την εφαρμογή και την εστρικοποίηση του εξωτερικού κόστου. Ήταν δύσκολη η αρχή. Ελπίζω όμως να σημειώσουμε πρόοδο προκειμένου να δώσουμε και ένα μήνυμα μέσω των τιμών για τη βελτιστοποίηση των μεταφορών και χρειάζονται και θέματα επιμελητίας και φιών τεχνολογιών. Γιατί θέλουμε να, είναι εφαρμόσιμα όσα αποφασίζουμε. Γιατί ξέρουμε ότι οι μεταφορές αποτελούν ένα μέσο για την ενιαία αγορά και αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες όπου μπορούμε να ενεργήσουμε πραγματικά. Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία σύντομη ερώτηση για τη μεθοδολογία. Στα στατιστικά σας στοιχεία, πώς λαμβάνετε υπόψη τις τεχνολογικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένους τρόπους μεταφοράς. Στις οδικές μεταφορές, για παράδειγμα, έγιναν πολλά για να γίνουν πιο αποδοτικά τα οχήματα από ενεργειακή άποψη. Έχει ε, μειωθεί αισθητά και ο αριθμός των σωματιδίων που εκπέμπονται από τα αυτοκίνητα. Εγώ είμαι Δανέζα, χώρα που ε, έχει την έδρα του ο οργανισμός. Και εκεί οι περιβαλλοντικές αρχές ισχυρίζονται ότι το καμποτάζ ε, ρηπαίνει πολύ περισσότερο το περιβάλλον από ό,τι οδικές μεταφορές. Και αυτό πραγματικά μας εξέπληξε. Και έτσι τέθηκε στη ημερήσια διάταξη και το θέμα των εκπομπών των πλοίων. Σε, άλλες, σε άλλους τρόπους μεταφοράς όμως, για παράδειγμα στις οδικές μεταφορές, εκεί οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι πιο αργές. Ε, και τα πλοία στη Δανία ρηπαίνουν, αλλά και τα τρένα, γιατί λειτουργούν με δίζελ και οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, δεν είναι αρκετά γρήγορες ώστε να αντισταθμίσουν το περιβαλλοντικό κόστος. Πώς λαμβάνετε υπόψη λοιπόν τις τεχνικές, τεχνολογικές αλλαγές στην έκθεσή σας όταν συγκρίνετε τους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Ο κύριος Σαβαρή. Σας ευχαριστώ. στις στατιστικές των μεταφορών και στην πολιτική των μεταφορών υπάρχει μια σταθερή. Εδώ και μία δεκαετία κάνουμε πολλές προσπάθειες προσώρες κατευθύνσεις για να χρησιμοποιήσουμε διαλειτουργικό τρόπο μεταφοράς και διατροπικό, ενώ σταθερά οι στατιστικές μας δείχνουν ότι ουσιαστικά διωγγώνονται οι οδικές μεταφορές και η αυτοκινητοβιομηχανία κερδίζει μερίδιο στην αγορά και στις μεταφορές προσώπων και στις μεταφορές εμπορευμάτων. Άρα κάπου πήγε στραβά η πολιτική μας, γιατί εδώ και μία δεκαετία προσπαθούμε με τον ΑΒ τρόπο να προωθήσουμε πιο φιλοπεριβαλλοντικές μεταφορές, πιο καθαρούς τρόπους μεταφοράς. Άρα θα πρέπει να καταλήξουμε στο σκληρό και το συμπέρασμα ότι δεν τα έχουμε καταφέρει. Εσείς ε, τι θεωρείτε ότι οι προσπάθειες ε, για διατροπικές ε, μεταφορές δεν είναι επαρκείς για να έχουν ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ή μήπως έχουν μόνο περιθωριακό χαρακτήρα. Και δεύτερη ερώτηση από όλη της πρώτης. Εδώ υπάρχει μια κατανομή αρμοδιοτήτων. Για τα βασικά στοιχεία όμως που άπτονται το πολιτικές μεταφορών, την αρμοδιότητα τη φέρουν άλλοι. Για παράδειγμα, για τα θέματα της έρευνας. Εγώ δεν γνωρίζω ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις. Γιατί είπατε ότι προβαίνετε σε συγκριτική μελέτη για το τι συμβαίνει. Ιδιαίτερα σε ό,τι φορά τους καθαρούς κινητήρες. Δεν νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον θα εγκαταλείψουμε τα ΙΟΤΑΧΗ. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν ε, προσπάθειες βελτίωσης μέσω όμως της ε, τεχνολογικής εξέλιξης. Ίσως δεν είναι η μόνη λύση, αλλά είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές. Εσείς έχετε κάποια μοντέλα στο μυαλό σας, ε, θεωρείτε ότι θα γίνει εξέλιξη τεχνολογική των οχημάτων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας ε, για απτές Βελτιώσει τεχνολογικές που αφορούν τους ίδιους κινητήρες, όχι θέματα λεπτομέρειες ραντάρ και την εκπομπή των ρήπων. Η κυρία Λίχτεμπεργκερ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το στατιστικό υλικό μπορεί να το δει κανεί με ψύχρεμο τρόπο και να εξαγάγει τα ανάλογα συμπεράσματα. Καταρχάς, οι εκπομπές αυξάνονται και ο ρυθμός ανάπτυξης δεν έχει περιοριστεί. Τώρα, επειδή αυτό δεν εμφανίστηκε στα στατιστικά στοιχεία, με την ενίσχυση, αν θέλετε, της ε, βιομηχανικής, ε, τη μείωση της βιομηχανικής ανάπτυξης, το διαπιστώνουμε αυτό όντως. Αλλά αυτό Προφανώς δηλαδή η μείωση των ε, ρήπων λόγω μείωσης ε, των ε, μεταφορών λόγω της ύφεση δεν αποτελεί φυσικά τον ευκταίο στόχο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεσή σας σε ό,τι αφορά την ανάγκη για τη διαχείριση της ζήτησης. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε τι βαθμό συμμετοχής ε, στις εργασίες για τα προϊόντα είναι απαραίτητος. Και αυτό είναι σημαντικό. Δεν βρισκόμαστε σε καθεστώς ε, δικτατορίας, θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ γεγονός, ότι είναι γεγονός ε, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αναφέρεστε στην προβληματική του PM10. Μειώνονται αυτές οι τιμές. Αλλά και πάλι είναι υπερβολικά υψηλές σε σχέση με τα επίπεδα που θα έπρεπε να είναι στις πόλεις. Κάποιες πόλεις οι οποίες ε, έχουν ε, καλούς ανέμους, είναι τυχερές, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε τα απαραίτητα μέτρα, ίσως να αλλάξουν και οι επιδοτήσει, για παράδειγμα, οι κανόνε για την επιδοτήση στον καυσίμων, γιατί είναι σημαντικό και αυτό. Τι μεταφορές θα πρέπει να κοιτάξουμε γενικά ότι δεν είναι η ποσότητα αυτή που είναι καθοριστική. Ή για παράδειγμα το γεγονός ότι λέμε μιλάμε για την οικονομία. Όχι, δεν είναι η ποσότητα, είναι η ποιότητα αυτή που έχει σημασία. Η ποιότητα είναι αυτή η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, για παράδειγμα και να κοιτάξουμε ποιο είναι το πιο σκόπιμο, ο πιο σκόπιμος στόχος. Επίσης είναι σημαντικό στο γεγονός ότι μιλάτε για την ενημέρωση των ε, επιβατών στον τομέα των δημόσιων ε, μεταφορών και εδώ θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά. Γιατί εγώ γενικά είμαι συνηθισμένη να χρησιμοποιώ τα μέσα μαζική κοινωνία, αλλά είναι πάντα δύσκολο αυτό σε ξένε πόλει. Να διαπιστώνουμε δηλαδή ε, που πάει, ποιο τρένο πάει πού, ποιο λεωφορείο πάει πού. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μα απασχολεί όλου. Χρειαζόμαστε καλύτερα συστήματα ενημέρωση. Αυτό αποτελεί την κατεξοχήν ε, πρόκληση για την τεχνολογία ενημέρωση. Αν το καταφέρουμε δε αυτό, τότε θα πείσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό με τρόπο φιλικό και προ του ηλικιωμένου. Για παράδειγμα, διαπιστώνω ότι οι ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, το συντρόδρομο ή τα λεωφορεία, γιατί ε, δεν ξέρουν πώ πρέπει να χειρίζονται τα μηχανήματα. Πολλέ φορέ έχω δει στην Αυστρία, στη Γερμανία, ε, ηλικιωμένου ανθρώπου να κάθονται και να κοιτάνε με αγορία τα μηχανήματα, γιατί δεν ξέρουν πώ να χτυπήσουν το στήριό του. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να ενημερώσουμε καλύτερα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο επηρεάζει πολύ την καθημερινή ζωή των οικογενειών για τη μεταφορά των παιδιών προς το σχολείο. ναι, αυτό είναι το σχόλιο για την οικονομική κρίση. Δεν ξέρω αν λέτε και τη σχετική έκφραση στα γερμανικά που λέμε στην Αυστρία με το κούκο. Η μεταφορά λοιπόν των παιδιών ε, προς το σχολείο. Γιατί όλο και πιο πολλοί γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους προς το σχολείο πρωτού πάνε στη δουλειά τους το πρωί. Και θεωρώ ότι πρόκειται για μία εξέλιξη η οποία δεν είναι ιδιαίτερα θετική γιατί καταρχάς τα παιδιά δεν ασκούνται ο βασικός λόγος που αναφέρεται είναι η ασφάλεια και ο φόβος των γονέων, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τελευταίο στοιχείο, η τεχνολογία. Σίγουρα δεν είναι η μοναδική οδός, αν θέλετε, για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά θα πρέπει να συμβάλλει και η έξυπνη τεχνολογία. Η μεταφορά δεν συνεπάγεται πάντα ευημερία, δεν υποφελούνται όλες οι περιφέρειες από την μεταφορά πολλές ε, περιοχές, πολλές περιφέρειες δεν εισπράττουν τίποτα παρά μόνο ζημιές από τις μεταφορές αυτές. Η κυρία Γελασέντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μακλέιτ για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης και έχω ορισμένες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Με ποιο τρόπο εντάσσει ο οργανισμός όλα αυτά τα μέτρα και τις αξιολογήσεις στο γενικό πλαίσιο των μεταφορών. Γιατί εμείς βλέπουμε τις στατιστικές για τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά και στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα. Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα γενικό πλαίσιο και σε αυτό το γενικό πλαίσιο λαμβάνουμε αποφάσεις, για παράδειγμα, για τη μείωση των εκπομπών ή των ρήπων των πλοίων. Και πολλές φορές δεν περιοριζόμαστε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν ο οργανισμός να εκτιμήσει την πρόοδο, γιατί όλο κακές ειδήσει ακούμε. Και από την συσσόρευση αυτή των κακών ειδήσεων αποθαρρύνεται ο τομέας αποκαρδιώνεται τελείως και αδρανεί. Υπάρχει μια ανισορροπία. Ω προ το γενικό πλαίσιο, την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εφαρμογή τεχνολογιών, μείωση εκπομπών και εφαρμογή νέων τρόπων ε, συνδυασμένων μεταφορών ε, θα πρέπει να υπάρχει, να συμπεριληφθεί στην έκθεση για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια κίνητρα στον τομέα για να προχωρήσει, να έχει ένα υπόδειγμα να μιμηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να περιλαμβάνονται και αυτά τα στοιχεία στην έκθεση. Τελευταία φαίνεται ότι οι εκπομπές ε, μειώνονται, ε, αυξάνονται λιγότερο από ό,τι το ΑΕΠ το τελευταίο καιρό. Ωραία, δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στι κακέ ειδήσει. Ωραία, να λέμε την πραγματικότητα, αλλά να δώσουμε και καμία θετική είδηση για να δώσουμε και ένα μήνυμα αισιοδοξία προ του μεταφορεί για να κινητοποιηθούν και να κάνουν κάποια επένδυση για να έχουμε και κάποια καλύτερη αποδοτικότητα των μεταφορών. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Πώς θα μπορέσει ο οργανισμός να βοηθήσει στην αξιολόγηση των προγνωστικών. Δηλαδή πώς θα θα μπορέσουμε να προβλέψουμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο περιβαλλοντικό πακέτο, για παράδειγμα, υπήρξε πρόταση για τη μείωση των ορυκτών καυσίμων μέσω πιο εκτεταμένης χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέχρι 10%. Και έγινε μια δημόσια συζήτηση, αλλά εκεί η επιλογή των βιοκαυσίμων προσέκρουσε στην ε, συζήτηση για την επιστηστική ασφάλεια. Και έτσι μπλοκαρίστηκε το θέμα των βιοκαυσίμων, που ήταν σημαντική εναλλακτική λύση σχέση με τα ορυκτά καύσιμα. Και με το θέμα της Ευρωβινιέτας. Εκεί πρότεινε αυτό το μέτρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση της συμφόρησης, αλλά την ώρα της αλήθειας διαπιστώσαμε ότι το μέτρο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας εξασφάλισε ουσιαστική μείωση των συμφορήσεων. Ερωτώ λοιπόν, με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την αξιολόγηση του οργανισμού που είναι πολύ αποτελεσματική και πώς μπορούμε το θέμα των συνδυασμένων μεταφορών, βελτίωση της ε, επιμελητίας, ε, διατροπικότητα, καλύτερη πλαισίωση της μετακίνησης ε, στις πόλεις, όλα αυτά τα στοιχεία πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν καλύτερα στη μελλοντική μας πολιτική για πιο αηφόρες μεταφορές. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς την εκπρόσωπο του Οργανισμού Περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά την ε, χωροταξία και την πολεοδομία. Πώς πιστεύετε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μεταφορές ε, σε αυτά τα πολεοδομικά σχέδια ή και στα χωροταξικά σχέδια. Θα πρέπει σίγουρα να ευνοήσουμε τις σιδηροδρομικές μεταφορές και δεν μιλώ μόνο για τις υπερταχίες, τα ΤΖΒ που αφορούν κυρίω τη μεταφορά επιβατών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε του σιδηροδρόμου, να βελτιώσουμε τι σιδηροδρομικέ υποδομέ ώστε στις ε, υπάρχουσες υποδομές ε, να κυκλοφορούν όλο και πιο γρήγορα τρένα. Εφόσον ε, οι υποδομέ είναι καλής ποιότητας, οι σιδηροδρομικέ μεταφορέ θα αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα θα πιστούν και οι επιβάτες να σε χρησιμοποιούν περισσότερο, γιατί θα πιστούν για την ε, αποτελεσματικότητά τους. Και οι πλωτές μεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές έχουν μεγάλο δυναμικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε τα λιμάνια του Δούναβη για παράδειγμα. Γιατί πραγματικά έχει τεράστιο δυναμικό ο Δούναβης και η εσωτερική πλωτή μεταφορά. Όπως και η περιοχή του Εύξηνου Πόντου. Ανεξάντλητο δυναμικό που μέχρι στιγμής μένει ανεκμετάλλευτο. Με τη διατροπικότητα πιστεύω ότι θα μειώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και σίγουρα χρειαζόμαστε φυση συστήματα μεταφορών, αλλά και να λάβουμε υπόψη και το θέμα της επιμελητίας, γιατί το θέμα των ε, ευφυών συστημάτων μεταφοράς και λογιστικά συστήματα καλής ποιότητας και αποτελεσματικά θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε και το χρόνο αναμονής αλλά και την ρήπαση που προκαλούν μεταφορές στο περιβάλλον. 10, Άντε δέκα λεπτά. Άλλα πέντε λεπτά. Για να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις στον χρόνο που έχω. Ξέρουμε ε, ποια άλλοι παράγοντες συμβάλλουν σε κομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και αν σας καθησυχάσω όσον αφορά τις επίκαιρες πληροφορίες. Τον επόμενο μήνα θα δώσουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και θα συμπεριληφθεί στην έκθεση που βληθεί στην ε, σύμβαση πλαίσιο του ΙΕ. Θα δούμε ποια είναι η συνεισφορά των μεταφορών και θα μπορέσουμε να δούμε και ποιες είναι οι συνέπειες της περσινής ημιύφεσης και της ε, οικονομικής κρίσης εκπομπές θα έχουν μειωθεί αναφυσβήτητα αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει αλλάξει συστημικά η εκπομπή αυτή. Λοιπόν, θα πρέπει να το παρακολουθούμε το θέμα. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι 40% της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας είναι στα νοικοκυριά. Πρέπει να παρακολουθούμε τα νοικοκυριά, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί και ο προβολέας πέφτει σε άλλες ε, ομάδες. Ας προχωρήσω όμως. Βεβαίως θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους σχετικά με την ανάγκη να ε, περιλαμβάνει να συγκρατήσει τις μεταφορές στο σύστημα εμπορίου ρήπων. Ε, θέλουμε να συμπεριληφθεί και οι διεθνείς, ε, οι διεθνείς αερομεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουν σε ένα γενικό πακέτο. Αυτό είναι σίγουρο και σε ελπίσουμε ότι καθοδόν προς την Κοπεχάγη θα μπορέσουμε να, να πείσουμε και άλλους συναδέλφους γι' αυτό. Υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί θαλάσσιες μεταφορές, η ναυσιπλοεία, η θαλάσσια, είτε είναι παράκτια ή γύρω στην Ευρώπη, στα πιο ανοιχτά, οι Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο είναι σε δύσκολη θέση γιατί πιέζονται να προτείνουν κάποιο πακέτο. Αλλά θα πρέπει πιο καταεπίχοντα και τα θιούχα και τα ζωτούχα να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, η θαλάσσια ναυσιπλοεία ε, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί. Είναι υπέρ της υγείας. Και χώρες όπως η Ολλανδία θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις επιταγές της νέας οδηγίας για τα ζωτούχα και για τα θιούχα που θα τεθούν αυτά σε ισχύ από το 2010. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί πολεμάνε οι χώρες με κάποια από τα σωματίδια, τα επίπεδα ε, PM10 και τα ζωτούχα το 2020 θα είναι μια πρόκληση. Ό,τι και να κάνουμε σίγουρα για τη θαλάσσια αναψυπλοεία θα βοηθήσουμε τις χώρες να ανταποκριθούν στις άλλες τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά τις συνέπειες στον τομέα του εμπορίου, δεν αναφέρομαι με κάποια σειρά προτεραιοτήτων στα θέματα, αλλά με τη σειρά υποβολή των ερωτήσεων. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα στην εσωτερική αγορά. Στο θέμα του καμποτάζου δεν έχουμε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, αλλά είναι σαφές ότι περίπου 1 με 10% απώλειες υπάρχουν ε, λόγω αδείων εμπορευματοκιβωτίων που πηγαίνουν δόθε και κήθε. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε το μεταφορικό σύστημα όσον αφορά την αποδοτικότητά του, ε, θα είναι καλό. Πρέπει να το κάνουμε αυτό που μπορεί να γίνει. Να μεταφέρει κανείς αέρα κοπανιστό, αέρα κοπανιστό σε κουτιά, δεν είναι κάτι αποτελεσματικό ίσως είναι, τι να πούμε, πιο καλός αέρας εδώ από ό,τι αλλού, αλλά τι να πω. Υπάρχουν κέρδη όσον αφορά την αποδοτικότητα. Μπορούμε παντού να κερδίσουμε. Λοιπόν, το μήνυμά μου που επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μία λύση. Κάθε κομμάτι του συστήματος θέλει επιδιορθώσεις και προσαρμογές και χρειάζεται τη δική μας προσοχή και την προσοχή της Επιτροπής σας. Όσον αφορά το εμπόριο, Απλώ η βελτίωση της εσωτερική αποδοτικότητας μετακινήσεως των εμπορευμάτων θα πρέπει να εξεταστεί η ποιότητα και η αποδοτικότητα των οχημάτων. Αυτό ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε για τα στοιχεία. Πάντα βλέπουμε τα πράγματα αναδρομικά. Άρα εξετάζουμε να δούμε την... τι γίνεται με τα κέρδη όσον αφορά την αποδοτικότητα. Και τα σχολιάζουμε. έχουμε διάφορες προδιαγραφέ ευρωπαϊκές. Προσπαθούμε να προβλέψουμε τι θα κάνουν τα μέτρα, μόνο αν εφαρμοστούν όμως βλέπουμε τα αποτελέσματα. Στην έκθεση σας δείχνουμε ιστορική εικόνα. Κατά πόσο η πρόοδο στην τεχνολογία έκανε κάποια διαφορά. Και όπως προανέφερα στην παρουσίασή μου, μπορούμε να ρυθμίσουμε τι γίνεται με τι εκπομπέ, τι βγαίνει από την εξάτμιση, αλλά αν κάποιο ε, θέλει να εμπλουτίσει το γιοταχή του με κλιματισμό κλπ, κλπ. Τι θα κάνουμε, που επιβαρύνει τι εκπομπέ. Έχω συζητήσει με του εκπροσώπου τη αυτοκινητοβιομηχανία. Και αυτό αφορά το μέλλον και τις πράσινες της απασχόλησης. Ποιο είναι το πρόβλημα σχετικά με την αυτοκινητοβιομηχανία και τους απασχολούμενους κατάντι ανάλογα με τη χώρα και τη βιομηχανία. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι ο τρόπος κατασκευής των αυτοκινήτων αφορά την ασφάλεια στους δρόμους. Οδηγούμε γρήγορα. Θέλουμε βαριά αυτοκίνητα για να μας προστατεύσουν σε περίπτωση σύγκρουσης. Αύξησε το βάρος των οχημάτων για να μας προστατεύει. Αυτό απαιτεί ατσάλι. Βαριά υλικά. Και κάποιες εταιρείες αλλάζουν τα υλικά τους. Υπάρχουν καινοτομίε όμως, έτοιμες να εφαρμοστούν. Ε, δεν έχουμε ε, πλαστικές καρέκλες στα αυτοκίνητα, καθίσματα στα αυτοκίνητα. Δεν είναι επειδή δεν δυνατόν αυτό, αλλά είναι διότι το εργατικό δυναμικό δεν είναι εκπαιδευμένο. Κάνουν ηλεκτροσυγκολήσει και ετοιμάζω τα οχήματα που έχουμε σήμερα. Δεν ξέρουν πώ να φτιάχνουν αυτοκίνητα από καλούπι. Στο πακέτο Ομπάμα βλέπετε ότι δίνονται χρήματα να καταρτιστεί ο κόσμο για να φτιάξει το αυτοκίνητο του μέλλοντος, αντί να χτίζει τα αυτοκίνητα του παρελθόντος. Άρα πρέπει να μάθουν να χειρίζονται νέα υλικά στο εργοστάσιο. Μην το ξεχνάμε αυτό όταν συζητάμε τα ευρωπαϊκά φορολογικά πακέτα και τις πράσινες θέσεις απασχόλησης και δημιουργία νέων δυνατοτήτων που δίνουν περιβαλλοντικά εφέλη αλλά αυτά τα μέτρα θα διατηρήσουν και τις θέσεις απασχόλησης και το εργατικό δυναμικό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν όσον αφορά τα στοιχεία και τα μοντέλα. Η υπηρεσία έχει στενότατα σχέση με τη Eurostat και άλλους φορείς και με τη βιομηχανία και πολλούς ομίλους μεταφορών. Έτσι συλλέγουμε πληροφορίες. Αλλά όλο και περισσότερο προσπαθούσαμε να βολιδοσκοπήσουμε το μέλλον, τι μορφή θα έχει και πώς θα εφαρμοστούν περιορισμοί περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αν θα πετύχουμε το στόχο του 2020, μηδενικές εκπομπές άνθρακα και σχετική οικονομία. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως για όλα αυτά. Ότι οι μεταφορές έρχονται πολύ πιο κάτω όσον αφορά τις εκπομπές αερίων. Πρώτος στόχος είναι η παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Μετά νοικοκυριά, σπίτια. Οι μεταφορέ είναι στην τρίτη-τέταρτη θέση. Μαζί με γεωργία, και ούτω καθεξής. Άρα δεν υπάρχουν κίνητρα για αλλαγέ να βάλουμε στόχο πενταετή, δεκαετή για μεταρρύθμιση του μεταφορικού τομέα. Και αυτό είναι το πρόβλημα όταν κοιτάμε το μέλλον. Ποιο θα έπρεπε να είναι, ποια θα είναι η μορφή της μελλοντική ε, μεταφορικής δομής. Περισσότερα ηλεκτρικά δίκτυα, περισσότερους, ε, περισσότερες διόδους ναυσιπλοείας, εσωτερικής ναυσιπλοείας κλπ. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη αρκετά στα διάφορα πακέτα πώς θα βοηθηθούν οι μεταφορές για να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Αν δείτε τι γίνεται στις χώρες, τι σχέδια έχουν, τι βλέπετε. Επικεντρώνονται στην παραγωγή ενέργειας κυρίως. Δεν επικεντρώνονται την προσοχή τους στις μεταφορές, εγώ έτσι τα βλέπω. Και σκεφτείτε το. Τέλο πάντων, τα πακέτα που υποβάλλονται τέτοια μορφή έχουν. Ποια είναι η απάντησή μου. Πρέπει να ξανασκεφτούμε το πώς θα προωθηθούν τα διάφορα πράσινα πακέτα. Και αν θέλουμε να πετύχουμε μείωση 80% αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, πρέπει να αλλάξουμε σημαντικά υποδομές. Η χρήση ανανοσίμων πηγών ενεργείας και τι γίνεται με την ηλεκτροδότηση, εξοικονόμηση τεχνικής ενέργειας, γλιτώνουμε μόλυνση, γλιτώνουμε θόρυβο και πιθανότατα πολλοί από εμά, λόγω της μολύνσης που αντιμετωπίζουμε, Ζούμε τουλάχιστον 8 μήνες λιγότερο. Μην πω, ακόμα λιγότερο. Σκληρά αυτά, αλλά αυτά κάνουν οι μεταφορές σήμερα. Δεν πρέπει να γίνονται έτσι όμως τα πράγματα. Ίσως να είναι τελευταία μου παρουσίαση σε αυτή την Επιτροπή και απευθύνω έκκληση. Μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά. Δεν χρειάζεται να έχουμε βαριά οχήματα που εκπέμπουν ρηπαντές στα κατόφλια μας και δεν χρειάζεται να γίνονται εκπομπές κοντά στα παιδιά μας. Σκεφτείτε το. Οι λύσεις υπάρχουν. Τα μοντέλα υπάρχουν. Είναι κάτι παραπάνω από πολιτική βούληση που χρειάζεται, αλλά η βιομηχανία, εάν ηγηθούμε, θα ακολουθήσει. Και η μεταφορά θα μπει στο εσωτερικό των πακέτων που αφορούν την ενέργεια και την καταπολέμηση αλλαγή του κλίματο. Αυτά και ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρο. Παρά το ότι αφιερώσα μόνο μία ώρα στο θέμα, έγινε πλούσια ανταλλαγή απόψεων, πολλά στοιχεία έχουμε, μπορούμε να τα σκεφτούμε είμαστε στο επίκεντρο των προβλημάτων στην επόμενη θητεία η Επιτροπή αυτή που ασχοληθεί με το θέμα είναι κάτι που κληροδοτούμε στο θεσμικό μας όργανο το οποίο θα συνεχίσει τη συνεργασία του. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που κάνατε μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα εξακολουθήσετε με αποτελεσματικό τρόπο και στο μέλλον έτσι. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Και είναι και το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων αυτής της Επιτροπής τουλάχιστον τυπικά, επίσημα, κανονικά αν και είναι αρκετά πιθανό αυτά που θα πούμε την επόμενη ώρα να μας υποχρεώσουν να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα τις επόμενες εβδομάδες στην Επιτροπή μας. Το θέμα είναι αυτή η κατανομή των διαφόρων σλότς και ανταλλαγή απόψεων. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της 16ης ε, Μαρτίου η Επιτροπή ήδη αντιμετώπισε αυτό το θέμα και αντιμετωπίζουμε πρόταση που υπευλήθη κατεπηγόντως ίσως ήταν υπερβολικά βιαστικές οι συνθήκες κυρίως διότι αφορά συμπεριφορές των αερομεταφορών από χθες, γιατί χθες την Κυριακή ξεκίνησε η θερινή εποχή 2009, η summer season, που αποτελεί αντικείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας που συζητούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε προσωρινή αναστολή λόγω της οικονομικής κρίσεως που περνάμε, αναστολή λέω, του κανόνα use or lose it, δηλαδή χρησιμοποιείς τη χρονοθυρίδα σου ή τη χάνεις, Επ, σας παρακαλώ. Μα, συγγνώμη, θα γίνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα αναστολή. Χρησιμοποίησε τη χρονοθυρίδα σου η Χάστιν, use it or lose it, που επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμά τους να διατηρήσουν αυτές τις χρονοθυρίδες, slots, όσοι έχουν δικαίωμα. Αν δεν καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν 80% τουλάχιστον αυτών. Αν κατά τη διάρκεια μέσα εποχής μια αεροπορική εταιρεία δεν χρησιμοποιεί το 80% των σλότ που προβλέπονται, το χάνει κανονικά. Αυτό πάει σε ένα εθνικό πουλ, σε εθνική ποσότητα, ποσόστοση που χρησιμοποιείται μετά. Ο λόγος αναστολής είναι η αντικειμενική οικονομική κρίση που αντιμετωπίζεται τώρα. Βρισκόμαστε μέσω κρίσεως, χωρίς να προβλέψουμε πότε θα βγούμε από αυτή την κρίση. Και η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι έλαβε και άλλες διφορές τέτοια μέτρα. 2001 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους και το 2003 όταν είχαμε την επιδημία ε, της SARS που ε, επηρέασε τις αερομεταφορές. Έχει δύο τμήματα η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπαμε έχουμε την αναστολή του κανόνα των διατάξεων από χθε μέχρι τέλος θερινής εποχής και μέχρι το 2010 μπορούν να χρησιμοποιούν τα slots που είχαν και πριν, ισχύσουν οι κανόνες και προτείνει μέσω ταχέστερης διαδικασίας από την επιτροπολογία με έλεγχο να μπορεί να χρησιμοποιεί την ίδια νομοθεσία για τη χειμερινή περίοδο. Αν διαπιστωθεί ότι συνεχίζεται η κρίση Αυτό είναι το ζουμί της πρότασης. Ήδη σαν Επιτροπή αποφασίσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την επιτάχυνση της διαδικασίας, διότι θέλουμε να κινηθούμε κατεπηγόντως, άρα θα εφαρμόσουμε τη διάταξη 43, δεύτερη παράγραφος, του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που πήραμε στις 16 Μαρτίου και αφού ακούσαμε και τα σχόλιά σας που μπορέσατε να τα σκεφτείτε και να τα αναλύσουμε όλα αυτά σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο αυτό θα πρέπει να συναγάγω συμπεράσματα από τη συζήτηση και τα συμπεράσματα αν είναι αναγκαίο να τα μεταφράσω, να τα μετατρέψω σε κάποιες τροπολογίες που θα προταθούν στον αφορά την πρώτη της και θα πρέπει να το κάνω αυτό ε, μέχρι το βράδυ. Θα πάρετε κάποια πρόταση μετά τη συζήτησή μας. Μετά τη συζήτηση σας κάνω εγώ προτάσεις. Τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το εσωτερικό κανονισμό έχουν 21 μέρες χρόνο και σε 21 μέρες αυτές. Αν δεν υπάρξει αντίδραση, άρα μέσω σιωπής σημαίνει ότι συμφωνείτε με την πρόταση, εν τη αυτή περιπτώσει η πρόταση υποβάλλεται αυτομάτως στην Ολομέλεια, εάν δεν γίνει αυτό, αν το 10% των μελών της Επιτροπής, δηλαδή 6 μέλη, μου γράψουν ότι δεν μπορούν να δεχθούν την πρότασή μου, αυτή η πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί σε ψηφοφορία στην Επιτροπή μας και μετά από αυτό αυτή η πρόταση Σύμφωνα το 43.2 περιορισμός είναι ότι οι τροπολογίες είναι αυτές που θα κάνω εγώ και καμία άλλη. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία θα ξαναρχίσει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτό σημαίνει Αν δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία επί μιας προτάσεως, επειδή υπάρχουν αποκλείωσες απόψεις στην Επιτροπή, προβλέπεται ψηφοφορία. Και προληπτικά ζητήσαμε να έχουμε σλότ και εμείς στην Ολομέλεια του Στρασβούργου 22 Απριλίου την 21η ημέρα, 22 του μηνός λοιπόν, θα πρέπει να συναντηθούμε, να συνεδριάσουμε σε ένα επιτροπή στο Στρασβούργο, εκτάκτος, ούτω ώστε ενδεχομένω να ψηφίσουμε την ελόγω πρόταση. 20, Δευτέρα, 22 Απριλίου, Στρασβούργο. Βεβαίως αυτή είναι διαδικασία συναπόφασης. Δεν ισχύει μόνο αυτό που κάνουμε εμείς αλλά επί οσδήποτε προτάσεως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου για να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αν δεν πετύχουμε συμφωνία μέχρι 5-6 Μαΐου στην πρώτη ανάγνωση, κλείνει το Κοινοβούλιο μετά και αναβάλλεται για την επόμενη θητεία το θέμα διότι θα πρέπει να πάρουν οι επόμενοι μετά την απόφαση. Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί και πιστεύω ότι με υποστηρίζετε να βρω μια λύση και να κάνουμε αυτό που γίνεται συνήθως. Μπορώ να σας πω ότι ήδη συμφωνούμε ούτως υπήν. Με την Τσεχική Προεδρία ανελήφθη υποχρέωση να τα πούμε μεθαύριο μετά τη συνεδρίασή μας. Χθες έγινε ανταλλαγή απόψε. Έχετε πληροφορήσει το Συμβούλιο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πολύ. Αρχίζω να ασχολούμαι ε, με το Συμβούλιο όταν βλέπω ότι έχει στα χέρια του το Κοινοβούλιο πρώτα. Θα πρέπει να συναντηθούμε με το Συμβούλιο, όμως μετά από το χρονικό διάστημα, κάποια λύση. Αυτή είναι η διαδικασία. Φαινόταν λογική και συνήθιση η πρόταση όταν κατέφτασε. Όμως τελικά απεδείχθη πιο περίπλοκη από ό,τι φάνηκε με πρώτη ματιά. Στι 10 μέρες ασχολούμαι με το θέμα. Προσπάθησα να καταλάβω κάποια πράγματα, τι απόψει του τομέα και θέλω να μοιραστώ μαζί σας εντυπώσεις που σχημάτισα. Και γι' αυτό ετοίμασα ένα μικρό έγγραφο που θα σα το μοιράσω όταν θα είναι έτοιμο, διότι οι ετοιμασίε γίνονται σε συνθήκες ιδιαίτερες. Τι διακυβεύεται όσον αφορά τα συμφέροντα. υπάρχουν διάφορα συμφέροντα θεμητά. Ποια είναι η καρδιά του προβλήματος. Έχουμε από τη μια τα συμφέροντα των network airlines, όπως αποκαλούνται, legacy airlines, των παραδοσιακών αεροπορικών εταιριών, που χειρίζονται τα δίκτυα πιο παλιές εταιρείες, όχι μόνο διαδρομές point to point, Τέλο πάντων, είναι αυτέ. Είναι incumbent. Είναι αυτέ που έχουν τι περισσότερε χρονοθυρίδε σε σχέση με τι άλλε εταιρείε. Αυτή είναι η πρώτη διάκριση. Αυτοί θεωρούν λοιπόν η καθιστική ατάξη των αεροπορικών εταιριών του ΣΥΠΗΝ βρίσκουν συμμάχους στα αεροδρόμια. Πριν από 10 χρόνια, πέντε χρόνια δεν ξέρω πόσα πριν, οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες υπήρχε, είχαν συσχετισμό με το αεροδρόμιο κόμβου με την αεροπορική εταιρεία. Air France ήταν Παρίσι, British Airways ήταν Heathrow κλπ. Συνδεόταν η μεγάλη εταιρεία με κάποιο αεροδρόμιο. Σήμερα όμως άλλαξε αυτό, δεν είναι πια έτσι. σχετίζεται εκεί που σχετίζεται το αεροδρόμιο με πιο πολλές από μία εταιρεία ε, έχει αδιαφορετική αντιμετώπιση από ότι μια συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Άλλαξε λοιπόν η γεωγραφική εικόνα. Λοιπόν έχουμε τις Network Airlines και την Non-Network Airlines, τις πιο καινούργιες. Έτσι γενικά. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους πελάτες, με τους επιβάτες. Οι επιβάτες ασχολούνται περισσότερο με το ποια, ποιος προορισμός κινδυνεύει. και δεν ξέρουμε κατά πόσο μέσω των νέων κανόνων κινδυνεύουν κάποιοι περιφερειακοί προορισμοί που, που εξυπηρετούνται από ρηπορικές εταιρείες μικρότερες και όχι τις network airlines. Ας πούμε εγώ έχω μια αεροπορική εταιρεία που έχω τα father rights, τα βασικά δικαιώματα. Και μου πούν το επόμενο εξάμεινο δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις χρονοθυρίδες όπως τα ήθελα και, διο, δεν σέβομαι τα όρια που έχουν καθοριστεί. Εγώ ήξερα ότι κινδυνεύω να χάσω τις χρονοθυρίδες, θα προσπαθούσα να, να προστατεύσω τα δικά μου, να μην έχω απώλειες, να μην έχω απώλεια κερδών, να χρησιμοποιήσω τις χρονοθυρίδες μου. Άρα, ίσως μπορεί μια... Ε, να μην εξυπηρετήσω μακρινό προορισμό και να, πάρω, να χρησιμοποιήσω το σλότ για πιο σημαντικό προορισμό. το δίκτυό μου το σχηματίζω όσον αφορά σε σχέση με, τις πιο, με τους πιο επικερδείς προορισμούς. Αλλάζουν οι προορισμοί έτσι. Και dalle compagnie aeree di network più remote sono quelle più a rischio. È più probabile che eh, come dire, l'esempio che abbiamo fatto le nostre discussioni con Air France era Συζητήσαμε και με την Air France. Διαδρομή Clermont-Ferrand Παρίσι δεν δεν θεωρήθηκε σαν μεγάλη, πολύ σημαντική διαδρομή. Δηλαδή, θα μπορούσε να κόψει αυτή τη διαδρομή αντί Παρίσι-Τόκιο, που είναι πιο επικερδής διαδρομή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το αντίθετο. Και αν δεν αναλάβει τη διαδρομή η μεγάλη εταιρεία, μπορεί να τρυπώσει η μικρή εταιρεία. Να αρπάξει σλότ τα οποία δεν μπορούσε να έχει πριν. Και μπορεί να τρυπώσει νέα εταιρεία. Αρκετά περίπλοκη κατάσταση όπως καταλαβαίνετε. Προσπαθούσα να τα δω όλα αυτά από αυτή την οπτική γωνία. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε σε κρίση, όχι μόνο τι αεροπορικές εταιρείε. και αεροπορικές εταιρείε έναν των άλλων φορέων των αερομεταφορών, αλλά να προστατεύσουμε και τους καταναλωτές και να επιβιώσουν οι υπηρεσίες από την κρίση. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις αεροπορικές εταιρείες, οι μεγάλες, οι network carriers, οι network airlines. Λένε ότι οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι σε δυσχερή θέση εναντί των υπολείπων αεροπορικών εταιριών. Διότι στη ΣΥΠΑ, η Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία επιδοτούνται. Ενώ εμείς δεν δεχόμαστε εθνικές χορηγήσεις. Και δεν τις βοηθάμε ούτε έμεσα. Αν εγώ πεινάω ας πούμε και μου δώσετε να φάω κάτι που μου κάνει δυσπεψία δεν είναι βοήθεια. Θέλουμε σωστή λύση. υπάρχει πρόβλημα ανταγωνισμού. Έχουν πρόβλημα οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έναντι των άλλων. Όπως είπα, τα αεροδρόμια βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Λένε, γιατί αν έχω μια εταιρεία που καλύπτει Παρίσι, Κλερμό, Φεράν, αυτή τη διαδρομή. Και Air France λέει, δεν θέλω να εξυπηρετήσω αυτή τη διαδρομή αυτό το δρομολόγιο. Σε αυτή τη διαδρομή, αν έχω waiting list και μου ζητάνε άλλοι χρονοθυρίδες, και δεν μπορώ να σου πω έχω ένα σλότ ελεύθερο. Εγώ λέω πάντα, εγώ τους έλεγα πριν πάντα όχι, γιατί μην τους πω ελάτε εσείς τώρα έχω χρόνο, αφού τον άφησε η Air France. Αν υπάρχει κρίση, η κρίση θα πλήξει όλες τις διαδρομές και διασυνδέσεις και δεν θα υπάρχει κανείς στην waiting list. Αν υπάρχει waiting list δεν υπάρχει κρίση. Άρα το αίτιο για το οποίο δεν μειώνονται πλέον τα slots Μάλλον η μείωση των χρονοθυρίδων είναι ανεξάρτητη από την οικονομική κρίση εφόσον περιμένουν οι άλλοι στην ουρά για να μπουν οι νέες αεροπορικές εταιρείες. Αν εγώ το αεροδρόμιο πρέπει να παρετηθώ από το να αντικαταστήσω την μεγάλη εταιρεία με κάποια άλλη εταιρεία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 Qual è la valutazione? Poi ho subito concluso. Λοιπόν, τελειώνω, τελειώνω. Τι γίνεται όσον αφορά τι Δεν υπάρχει αμφιβολία, υπάρχει κρίση. Διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει τώρα η κρίση από το 2001 και το 2003. Δεν αφορά μόνο την, ε, τις αερομεταφορές, δεν είναι aviation specific, αφορά όλους. Δεν μπορούμε να σώσουμε ένα τομέα βάρος άλλου διότι και άλλος τομέας αντιμετωπίζει κρίση. Πώς να το πω τώρα. Το 2001 και 2003 μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον υπόλοιπο κόσμο να βοηθήσει τον τομέα που επλήτεται από την κρίση δίδυμους πύργους ή SARS. Σήμερα πρέπει να προσέξουμε πώς παρεμβαίνουμε για να μην μεταθέσουμε το βάρος της κρίσης μην υποστούν τα αεροδρόμια τελικά αυτό που δεν θα υποστούν οι αεροπορικές εταιρείες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε την κρίση. Πριν ξέραμε ότι είναι προσωρινό πρόβλημα, μπορούσε να παρέμβει κανείς για ένα εξάμεινο και τελείωσε. Εδώ μπορεί να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε και εφόσον δεν ξέρουμε πότε θα λήξει η κρίση, δεν ξέρουμε πότε θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Άρα, μπορεί να διακόψουμε, να παρέμβουμε, να αλλάξουμε, να επηρεάσουμε την κίνηση σε αυτό τον τομέα για κάτι απρόβλεπτο. Δυστυχώς, τρίτον, επιτίθεται, αν θέλετε, επικάθεται η παγκόσμια κρίση επιτομεακών κρίσεων, απομονωμένων. Υπάρχουν αεροπορικές εταιρείε που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες από άλλες και για τις οποίες χρειάζεται αναδιάθρωση πλήρης αυτός εδώ, αυτή, αυτή η νομοθεσία θα μπλοκάριζε τη διαδικασία αναθεώρησης και αναδιάθρωσης. Συνοπτικά. Τελικά. Νομίζω πρέπει να προσέξουμε και τη λύση που θα δώσουμε. Και επιμένω ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τις μεγάλες εταιρείες, τους major stakeholders, αλλά τους τελικούς καταναλωτές, τους επιβάτες που ίσως να πληγούν Πρέπει να θυμόμαστε. Ότι μπορούμε να, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο των slots μόνο αν δεν υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να εργαστούμε σε πολλαπλά μέτωπα. Διερωτώ, διερωτάμε, διερωτώμε μας, συγγνώμη. Μήπως να μην είμαστε τόσο ομιμήσως να μπορούμε να διευκολύνουμε το σεβασμό των κανόνων, να σέβονται οι αεροπορικές εταιρείες τους κανόνες. Να αλλάξουμε κάπως την κατανομή των χρονοθυρίδων 75-25, ε, 70-30. Να λάβουμε κάποια μέτρα που λαμβάνουν υπόψη την κρίση. Να δεχθούμε μία μείωση που δεν είναι γενικής φύσεως αλλά να είναι μια αλλαγή η οποία να αναλογεί στην κρίση που αντιμετωπίζεται. Όσον αφορά τους επιβάτες, μετά πρέπει να βρούμε λύσεις που προστατεύουν το συγκεκριμένο τομέα. Ας πούμε, αν η Ελιτάλια πει δεν κάνω Παρίσι, Κλερμον Φεράν ή Air France. Θα πρέπει όμως να, να, να εκτελείται το δρομολόγιο Παρίσι, Κλερμον και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο, αν φύγει μεγάλη εταιρεία, να μην κάνει ότι του κατέβει, να το ξαναπώ, διευκολύνουμε τους κανόνες να συμμορφωθούν οι incumbent. Διευκολύνω να μπορούν να πούν οι νέες εταιρείε όσες θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα slot. Και να κάνουν όμως αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή που δεν καλύπτεται. Να βρούμε πώς μπορούμε να συγκεράσουμε τα διάφορα συμφέροντα. Διότι διαφορετικά με ομόν τρόπο θα πρέπει να μεροληπτήσουμε. Βλέπω ότι ο κ. θα έφεσε στα όρια της υπομονής του. Σταματώ εδώ και του δίνω το λόγο. Ο κ. Ζεμπόφσκι λοιπόν έχει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε, αναφέρατε τα πολλαπλά συμφέροντα που υπάρχουν εδώ στο παιχνίδι μεταξύ της μίας ε, αεροπορικής ε, εταιρείας, των αεροδρομίων, των επιβατών, Τόσο καλά τα είπατε όλα που δεν χρειάζεται καν να σχολιάσω. Θα ήθελα να παρουσιάσω την θέση του ΕΛΚ κατά πλειοψηφία, κατά την εξέταση των ξεχωριστών συμφερόντων και επειδή μιλάμε για μία σεζόν θεωρούμε, δηλαδή δεν θα συμφωνήσουμε με την πρόταση παριθμών 3 για την ε, αόριστη επιμήκυνση παράταση του μέτρου αυτού μέσω επιτροπολογία. Μιλάμε για μία σεζόν. Θεωρούμε λοιπόν, θεωρεί το ΕΛΚ ότι λόγω της βαθιάς κρίσης που έχει πλήξει την Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάναμε πάρα πολύ καλές συζητήσεις μαζί σας και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Νομίζω ότι οι αλλαγές για το 80, 20, 70, 30 δεν έχουν ε, πολλά να προσφέρουν. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θέλουμε για έξι μήνες να είναι σαφής η θέση μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρη η θέση του ΕΛΚ. Θα ανακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μεταξύ άλλων επειδή αυτό αποτελεί και την άποψη της πλειοψηφίας του Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, το τονίζω αυτό. Αν ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή για 6 μήνες θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα την όλη διαδικασία γιατί θέλουν και μία απάντηση, σαφή απάντηση. Οι αρεολιμένες δεν θέλουν να μπλέξουν στην όλη διαδικασία της επιτροπολογίας. Δεν αξίζει τον κόπο για 6 μήνες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρεί η ομάδα μου ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 10C 10C1 και 2 και να καταψηφίσουμε την πρόταση υπαριθμών 3. Αυτή είναι η άποψή μου, η δική μου και η άποψη της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Well, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λίγο πριν από μία εβδομάδα θα μπορούσα να σα είχα μεταφέρει την γνώμη της ομάδας, αλλά στο μεταξύ φαίνεται ότι υπάρχουν αλλαγές. Θα δώσω την προσωπική μου άποψη μόνο. Την περασμένη εβδομάδα, όταν συζητήσαμε το θέμα, νόμιζα ότι η ομάδα μου θα σας υποστήριζε. Αλλά η κατάσταση τώρα έχει αλλάξει, άρδιν. Υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις τις τελευταίες τρεις-τέσσερις μέρες και η ομάδα μου έχει αλλάξει γνώμη. Τώρα ο Γιώργ λέει ότι το έλκυν υπέρ της αναστολής του κανονισμού για τα σλότ, για τις χρονοθυρίδες. Ουσιαστικά είστε υπέρ της εγκατάλειψης των δυνάμεων της αγοράς. Ενώ για 20 χρόνια μας έκανε κήρυγμα για το πώς η απελευθέρωση της αεροπορίας είναι ο καλύτερος τρόπος, πώς θα πρέπει να αφήσουμε την αγορά ελεύθερη. Αυτά δεν μας έκανε 20 χρόνια, Γκέοργ. Δεν ξέρω <laughs> Είσαι φάουλ τελείω. Δεν ξέρω αν γνωρίζει την ορολογία του ποδοσφαίρου, αλλά είσαι τελείω φάουλ. Μα αυτό είναι στρέβλωση της αγοράς. Είναι στρέβλωση της αγοράς που ασκείται από ορισμένε αεροπορικέ εταιρείε που ασκούν πίεση στις κυβερνήσεις του στις χώρες τους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί αυτό το επιχείρημα. Καλά, εγώ σα λέω την άποψή μου. Πάντως, εγκαταλείπουμε ή μάλλον αναστέλουμε τις ε, πρακτικές της απελευθερωμένης αγοράς ενδίδοντας ε, τον προστατευτισμό που μας ζητούν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες. Δεν θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Τι θα πρέπει, να αναστείλουμε όλες τις μορφές απελευθέρωσης. Να αναστείλουμε και την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, για παράδειγμα. Γιατί όχι, μπορεί και εκεί να επικαλεστείτε το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης γιατί δηλαδή οι αεροπορικές εταιρείες είναι διαφορετικές από τους άλλους κλάδους και αξίζουν αναστολής. Και άλλοι κλάδοι μαστίζονται από την οικονομική κρίση. Όλοι υφίστανται την κρίση. Γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε ειδικά τις αεροπορικές εταιρείες και όχι τα αεροδρόμια. Γιατί να υποστηρίξουμε τα, τις αεροπορικές και όχι τα ταχυδρομεία για παράδειγμα, όχι τους παραγωγούς ενέργειας, όχι τους σιδηροδρόμους. Πιστεύω ότι η αναστολή θα στρεβλώσει την αγορά της, ε, των αερομεταφορών, θα περιορίσει τι νέες εισόδους και θα εμποδίσει τις άλλες εταιρείες να, χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιεί τα σλότ. Έρχονται οι αεροπορικές εταιρείες, μας λένε αντιμετωπίζουμε κρίση, κρίση βοηθήστε μας, αλλά τα σλότ τα θέλουμε. Απλώς θέλουμε εσείς να μας κρατήσετε και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Ο πρόεδρος επισήμανε τα αποτελέσματα που θα έχει ένα τέτοιο μέτρο, ιδιαίτερα στα περιφερειακά αεροδρόμια. Γιατί οι πρώτες χρονοθυρίδες που θα έχουμε δεν θα είναι Παρίσι-Τόκιο, δεν θα είναι γραμμή Λονδίνο-Νέα Υόρκη. Οι πρώτες χρονοθυρίδες που θα φύγουν θα είναι προς τα περιφερειακά σας αεροδρόμια. Σε αυτά τα καημένα τα, τα περιφερειακά αεροδρόμια. Μην έχετε ψευδεστήσει. Και για το κατά πόσο η οικονομική κατάσταση για αεροπορικέ εταιρείε είναι τόσο δεινή όσο ισχυρίζονται, πολύ αφιβάλλω. Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε εγγυήσει και να σώσουμε για ένα εξάμεινο τι αεροπορικέ εταιρείε, όχι λόγω τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά επειδή το καπιταλιστικό σύστημα τη αγορά έχει καταρρεύσει και ξαναγκάζει τι εθνικέ αεροπορικέ εταιρείε να ζητούν κρατική προστασία. Η οικονομική κατάσταση είναι τόσο σοβαρή για, τις, για ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, κύριε Πρόεδρε, που έχουν τρελαθεί να αγοράζουν άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό είναι, αυτή είναι η έννοια της κρίσης. Ενώ υποτίθεται ότι πίσω κρίσης πέφτουν να αγοράσουν άλλες αεροπορικές εταιρείες. Δεν έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το χρήση στέρηση, το use it or lose it. Θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες εναλλακτικέ λύσεις. Για παράδειγμα, αν η πρότασή σας δεν συγκεντρώσει πλειοψηφία, πιστεύω ότι θα πρέπει να θέσουμε πολύ σοβαρές προϋποθέσεις, πολύ αυστηρούς όρους, που ούτως ή άλλως κατά τη γνώμη μου χρειάζονται. Εγώ επι επιμένω αναστολή να γίνει άπαξ και να μην επαναληφθεί μετά από δύο χρόνια. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει «Α, δώστε μας την εξουσία να μπορούμε να παρατείνουμε για άλλο ένα εξάμεινο και πάλι μέσω της επιτροπολογίας». Φυσικά, εγώ συμφωνώ με την πρότασή σου ότι δεν θα το δεχτούμε κάτι τέτοιο, αλλά αν αρχίσει τέτοια παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πάει εκείνη σε ευρωεκλογές ε, του Ιουνίου. Νομίζω ότι έχουμε τώρα την ευκαιρία για μια πλήρη αναθεώρηση του συστήματος των χρονοθυρίδων προκειμένου να υποβληθεί μια νέα πρόταση για να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι όσοι έδωσαν τη γνώμη τους λένε ότι το σύστημα χρειάζεται τροποποίηση. άκουσε ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει. Πού είναι η συμφωνία, το ακόμη δεν έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο. Εγώ από βολιδοσκοπήσεις που ειναι η συμφωνια το ακομη δεν εχει συμφωνησει το συμβουλιο εγω απο βολιδοσκοπη που εκανα για να μάθω τη θέση του Συμβουλίου είναι ότι μέχρι στιγμή έχει γίνει απλώς συζήτηση προσανατολισμού στο Συμβούλιο και ορισμένε χώρε, για παράδειγμα οι σκανδιναβικέ, οι είναι κατά τη αναστολή τη ρήτρα χρήση υστέρηση, use it or lose it. Δεν είναι λοιπόν δεδομένο ότι θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. Η πρόταση της αναστολής της ρήτρα αυτής έχει γίνει μόνο και μόνο για να καθησυχαστούν, κατευναστούν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εις βάρος της πολιτικής αεροπορίας γενικώ και εις βάρος του επιβατικού κοινού. Ευτυχώς ε, σε μία ώρα θα τελειώσει η συνεδρίασή μας και θα πρέπει να σε ξαναυποστούμε Γεώργο, όσο σύντομος και αν είσαι. Νομίζω δεν είναι αυτή η καλύτερη λύση. Αν θέλουμε λύση, θα πρέπει να βρούμε λύση για το σύνολο τη πολιτική αεροπορία και όχι μόνο προ όφελο ορισμένων αεροπορικών εταιριών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στέρξ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει γίνει αυτή η συζήτηση και έχει ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι και σε άλλες ομάδες θα πρέπει να συνεχίσουν οι συζητήσεις. Και εμεί δηλαδή στη δική μα ομάδα έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει ακόμα να τα εξετάσουμε. Αλλά νομίζω, Πρόεδρε, ότι αυτό που λέει ο Μπράιν Σίμψον δεν σύμφωνα απόλυτα μαζί του όταν ε, φάβει τον καπιταλισμό, αλλά συμφωνώ μαζί του όταν λέει ότι η γραμμή που ακολουθούμε είναι μια αρκετά λογική γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Ευσεβή πόθη, Μπράιαν. Υπάρχουν πολλά αντιφατικά συμφέροντα. Μια αγορά η οποία έχει απορριθμιστεί. Δεν βλέπω να υπάρχει όμως κρίση την οποία να θεωρούμε με, με στοιχεία ότι θα είναι βραχυπρόθεσμη. Και δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τα αεροδρόμια να προβούν σε τέτοια μέτρα. Μπορούμε να συζητήσουμε, Πρόεδρε, τα ποσοστά, αν θέλετε, αν θέλετε να χαμηλώσουμε, να αυξήσουμε τα ποσοστά 70%, 75%. Αλλά νομίζω ότι η γραμμή που ακολουθείτε και λέτε, δηλαδή, ας ε, περιορίσουμε το θέμα, ας περιορίσουμε τα ποσοστά και να δούμε εφόσον χρησιμοποιεί κανείς ένα σλότ να υπάρχει εγγύηση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Να εξασφαλίζεται δηλαδή η παροχή της υπηρεσίας για κάποιο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η γραμμή, αλλά δεν έχει υποθεί ακόμα η τελική αυτή λέξη αν θέλετε. Και έχουμε πολλά να συζητήσουμε και εμείς στην ομάδα μας και σε άλλες ομάδες. Ο κ. Αλμπερτίνη. Presidente, eh, la tua esposizione iniziale è stata esaustiva. Εξαντλητική και πλήρη η αρχική σα παρουσίαση, Πρόεδρε, και νομίζω ότι επαρκώ ε, παρουσιάζει τα στοιχεία. Συμφωνώ με το συντονιστή. Χρειάζεται αυτό το νομοθέτημα για την αναθεώρηση του κανονισμού 12593. Όμω, πιστεύω ότι χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ιδιαιτερότητες, κάποιες ιδιαιτερότητες που άπτονται όλου του τομέα των αερομεταφορών, όχι μόνο τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά όπως υπεθυμίστηκε και τα αεροδρόμια. Η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια πράγματι και γενική, πλήττει όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία και όχι μόνο τομέα συγκεκριμένο. Και ίσως αυτή η αναστολή του μέτρου θα πρέπει να εξεταστεί ως ενδεχόμενο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις, να πω σε κάποιες λεπτομέρειες, να αποσαφηνίσω. Υπάρχουν κάποια αεροδρόμια. Εκεί δεν υπάρχει κρίση όσον αφορά τη ζήτηση, αλλά κρίση προσφοράς. Εξηγούμε. Σε κάποια αεροδρόμια της πόλης μου, στο Λινάτε και στο Μαλπένσα, ο η βασική αεροπορική εταιρεία αλλά μεταθέτει το δίκτυο για βιομηχανική στρατηγική. Και η προσφορά μειώνεται λόγω αερομεταφορέα, όχι λόγω δυνάμεων της αγοράς και ζήτησης. Αυτό αφορά και άλλα αεροδρομία στην Ευρώπη. Θα υπήρχε λοιπόν ζήτηση, αλλά δεν θα καλυπτόταν λόγω ελήψεως οργανωτικής δομής από πλευράς του αερομεταφορέα. Υπάρχουν και αεροδρόμια που υπόκειται σε περιορισμούς λόγω του δυναμικού τους, των δυνατοτήτων τους για λόγους ασφαλείας και άλλα αεροδρόμια point to point που δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, για να σώσουμε την αρχή του ανταγωνισμού που είναι κριτήριο αποδοτικότητας της αγοράς που πρέπει να διαφυλαχθεί. Και για να γίνει παρέμβαση στην οικονομική κρίση θα έπρεπε ίσως να λάβουμε υπόψη την αναστολή μόνο στα αεροδρόμια εκείνα των οποίων έχει πληρωθεί το δυναμικό. Δεν έχουν άλλες δυνατότητες να καλύψουν τη ζήτηση. Και ίσως θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε το άρθρο 10, παράγραφος 4 που ξέρει ο Πρόεδρος. Τέσσερις γραμμές για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφους 4 οι συντονιστές των αεροδρομίων έχουν την, που έχουν εκπληρώσει το δυναμικό τους ε, θα αναγνωρίσουν ότι σε αυτά τα αεροδρόμια αεροπορικές εταιρείες κατά τη διάρκεια την περίοδο προγραμματισμού του καλοκαιριού του 2010 να έχουν τις ίδιες χρονοθυρίδες που τους είχαν ανατεθεί κατά το καλοκαίρι του 2009. Έτσι διαφυλάσσεται η αρχή της προστασίας των συνθήκων στους οποίους κινούνται οι αερομεταφορείς και θα μπορούν και οι επιβάτες να έχουν προσφορά, να έχουν υπηρεσίες και δεν πλήττονται και τα αεροδρόμια. διότι λόγω της ε, αναστολής αυτού του μέτρου ενδεχομένω να μειωνόταν σημαντικά η ζήτηση σε συγκεκριμένα αεροδρόμια και να αντιμετώπιζαν προβλήματα. Ο κύριος Στόκμαν, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είχα καταρτήσει τον κανονισμό για τα Σλότ και είχα λάβει εξαίρεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ με την ε, πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δυστυχώ να σα πω ότι δεν συμφωνώ με την προσέγγισή σα Και να πω και γιατί καταρχά ε, από πλευρά πολιτική μεταφορών. Έχουμε κάποια συμφέροντα τα οποία είναι σαφή. Υπάρχει μια έντονη κρίση και θέλουμε στην κρίση αυτή να μην γίνονται οικολογικές και οικονομικές ανοησίες. Και αυτό ακριβώς γίνεται όταν οι αεροπορικές εταιρείες να θέσω έναν όρο όμως ε, που δεν έχει τεθεί. Έχουμε μια νομισματική αξία για τα σλότς, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, διώκει πλέον την εμπορία των σλότς. Έχουν δηλαδή ε, μια νομισματική αξία που μπορεί να εξωτερικοποιηθεί. Δηλαδή, καμία αεροπορική εταιρεία δεν θα αφήσει εθελοντικά, αν θέλετε, ή θελημένα ένα σλότ. Θα το πουλήσει αν χρειαστεί για τον κανονισμό το 80 και 20. Μπορεί να χρησιμοποιούνται μικρότερα αεροσκάφη, αλλά όχι άδεια. Θα προσπαθήσουν δηλαδή να τηρήσουν αυτούς τους κανονισμούς. Αυτό είναι οικολογική και οικονομική ανοησία σε μια τέτοια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και πρόκειται για μια βαθιά κρίση που μας μαστίζει. Γιατί είναι σωστή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναστέλει τη ρύθμιση αυτή προκειμένου να σταθεροποιηθεί η αγορά, όχι να αποσταθεροποιηθεί και τελικά υποφέρουν μικρές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες οικονομικά είναι υποπίεση. Όχι οι μεγάλες, οι μεγάλες θα επιβιώσουν την κρίση φυσικά. Η πρότασή σας φαίνεται αρχικά ότι έχει καλές προθέσεις. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι μια ευελιξία στο όλο σχέδιο, αλλά νομίζω ότι ελοχεύει ο εξή κίνδυνος. Ανοίγουμε ένα νέο μοντέλο. Είναι μοναδική η κατάσταση, σας το λέω και για αυτές τις μοναδικές ε, καταστάσεις όπως το ΣΑΡΣ 11 Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα μοντέλο. Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι μοναδική αυτή η κατάσταση θα ξεκινήσουμε μια συζήτηση η οποία θα ανοίγει σε κάθε περίπτωση. Μήπως για κάθε περίπτωση οικονομικής κρίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτόν τον κανόνα το 80-20. Αυτό είναι λάθος. Είναι ένα πολιτικό βήμα, ένα πολιτικό εμπόδιο αν θέλετε. Το ταμπού αυτό θα πρέπει να διατηρήσουμε και θα πρέπει να το αφήσουμε και για τα φορτηγά, να μην το συζητάμε δηλαδή ξανά και ξανά, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν βοηθούμε και τους αερολιμένες. Νομίζω ότι δεν έχουμε κατανοήσει, δεν έχετε κατανοήσει τι θα πετύχετε αν περάσει αυτή η παράδοξη ρύθμιση. Άρα εγώ είμαι υπέρ της πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να περιπλέξουμε υπερβολικά ε, τη συζήτηση μιλάμε για έξι μήνες και ναι συμφωνώ να μην υπάρχει αυτόματη ανανέωση αλλά να μην θέσουμε και προς συζήτηση ένα νέο μοντέλο το οποίο δεν ξέρουμε τι θα συνεπάγεται για το μέλλον. Κοιτάξτε μια διευκρίνηση. Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για εξάμεινο. Πρόκειται για έξι μήνες από τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή συζητάμε τουλάχιστον για ένα χρόνο φανταζόμενοι ότι δεν ισχύει για το δεύτερο εξάμεινο και φτάνουμε το 2011. Χρονικό όριο δεν υπάρχει. Για ένα χρόνο μιλάμε. Ένα εξάμεινο και το εγγυόμεθα και τον επόμενο χρόνο. Πρώτη συνέπεια. Δεν παρεμβαίνουμε για να αλλάξουμε τη ισορροπία της αγοράς. Εάν δεν θέλουμε να κάνουμε καμία παρέμβαση θα αποσύρουμε το μέτρο. Δεν τίθεται έτσι το θέμα. Κύριος κύριε Γιαζεμπόφσκι, είμαι πολύ υπομονετικός, όμως αρχίζω, αρχίζει κάπως να εξαντλείται η υπομονή μου ε, έναντι τέτοιων σχολείων. Αν έχετε να πείτε κάτι, σηκώστε το χέρι να μου το πείτε, αλλά έτσι, αού, διάφορες φωνές κλπ. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύρκοπ έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα επανέλθω στο θέμα που συζητείτε το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι τα σχόλια του Μπράιν είναι πολύ παράξενα όταν προέρχονται από εκπρόσωπο της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου που τυπώνει και ε, ρίχνει χρήματα στην αγορά σαν να μην υπάρχει επαύριο. Κάτι τέτοιο τόσο πρακτικό που εξετάζει η Επιτροπή, η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή αντίθεση σε αυτή την απίστευτη, ανεύθυνη ε, και παρορμητική δράση της Βρετανικής κυβερνήσεως. Ο Τζορτζ Γιαζεμπόφσκι αναφέρθηκε Μπράιν στη Γενική Αρχή και πήρε απάντηση όσον αφορά τον Τζορτζ Γιαζεμπόφσκι και ότι δεν χρειάζεται να τον εκθεί άλλο, νομίζω ότι θα χάσει πολλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα είναι εδώ, Τζορτζ. Δεν είναι μόνο δική μου άποψη, αλλά τη πλειοψηφία τη Επιτροπή υποψιάζομαι. Γεγονό, Πρόεδρε, όσον αφορά τα θέματα που συζητούμε. Δεν θέλουμε να σε διακόπτουμε πολύ, Μπραάμ. Μην με διακόψει και εσύ τώρα. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Έχουμε σοβαρή οικονομική ύφεση. Πλήττει σκληρά ε, τι αερομεταφορέ και θα πρέπει να λάβουμε κάποια μέτρα αν μπορούμε. Όπω τα βλέπω εγώ και οι συνάδελφοί μου, εγώ υποστηρίζω με δισταγμό να παγώσει ο κανονε 80 80-20, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί το μέτρο και να μην ξεπεράσει το χρονικό όριο του Οκτωβρίου και να προκαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο. Τώρα θα προτείνει μια αναθεώρηση οδηγία για την κατανομή των χρονοθυρίδων. Εμείς το ζητούσαμε επί μακρόν. Είναι απαραίτητο. Και είναι ευκαιρία τώρα να προτείνουν κάτι. Και η αδίποτα αναθεώρηση δίνει έξοχη δυνατότητα θέσπισης μέτρων για οικονομικές κρίσεις και στο μέλλον. Και αυτή είναι μια δυνατότητα που θα πρέπει να αρπάξει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, να δουν και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι χειριστές των αεροδρομίων, οι συντονιστές των αεροδρομίων. Αντιμετωπίζονται προβλήματα στα αεροδρόμια, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Συστήνω πρώτα απ' όλα μια επανεξέταση των κανονισμών περί αεροδρομίων, ποιο είναι αντίκτοπο τη οδηγία για τα τέλη αεροδρομίων που καλύπτει τα μεγαλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη, πρέπει να αναθεωρηθεί. Μπορούν να γίνουν αλλαγέ επίση προσωρινά ή αναγκαίων ούτω ώστε να μην υποφέρουν επιβολικέ ρυθμίσει στα αεροδρόμια. Οι κανονισμοί αεροδρομίων θα πρέπει να έχουν, δίνουν κίνητρα οικονομικά ε, σε μικρά αεροδρόμια και να δίνεται και βοήθεια για να μπορούν να ξεκινούν αεροδρόμια. Η ασφάλεια των αεροδρομίων πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι χρηματοδοτείται από τα δημόσια ταμεία. Χρειάζονται εγγύησει από το Συμβούλιο ότι πραγματικά θα εξετάσει το θέμα, θα το συζητήσει το ταχύτερο δυνατόν οι εθνικοί φόροι αερομεταφορών πρέπει να εξαλειφθούν και θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία Ευρωπαϊκής ή των χωρών. Ε, κατεπηγόντως, αυτό θα έχει αντίκτυπο όσον αφορά την ασφάλεια και το γενικό κόστος που αντιμετωπίζει ο τομέας. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει κάποιες θετικές απαντήσεις όσον αφορά τις δυνατότητες που θίγω, εγώ πρώτος απ' όλους θα υποστήριζα το μέτρο που μας προτείνουν. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Οι αερομεταφορές, όπως είπε και ο Μπράιαν, είναι περίπλοκος τομέας. Πάντα υπάρχουν διασυνδέσεις και αντίκτυποι. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτό το πάγωμα, την αναστολή, για όνομα του Θεού, εξετάσουμε κάποιου τομεί και ιδιαίτερα τα αεροδρόμια και α του δώσουμε και εκεί χείραν βοηθεία στη δύσκολη εποχή που περνούν. Ε, bon, Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με αυτά που είπε ο Μπράιν Σίμψον, γιατί βλέπουμε εδώ εξόφθαλμες αντιφάσεις σε σχέση με αυτά που μας λέγατε πριν από 10 χρόνια για την απελευθέρωση των σλότ και των αγορών και τώρα την ανάγκη να παγιωθεί μια κατάσταση. Αλλά εδώ δεν είμαστε G20, άλλοι ε, είναι αρμόδιοι για την αναμόρφωση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. Ε, εγώ θα σχολιάσω λίγο τις δυσκολίες ε, του αεροπορικού τομέα. Πραγματικά σε τρεις μέρες η κατάσταση άρδεξε άρδια στους σοσιαλιστές, μας το είπε ο Μπράιαν, γιατί όλοι ζητήσαμε πληροφορίες και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μείωση των αερομεταφορών. Και από γαλλικές πηγές, δεν ξέρω αν είναι οικουμενικές ισχύω οι πληροφορίες, πάντως οι προβλέψεις μας για τις θερινές διακοπές ε, δείχνουν ιστορική χαρακτήρα μειώσεις ε, σε ό,τι αφορά την, ε, τις καλοκαιρινές διακοπές. Πραγματικά άνευ προηγουμένου η μείωση των ε, ταξιδιών των καλοκαιρινών. Οπότε ρεαλιστικά προσπαθούμε να σώσουμε τις αερομεταφορές όπω όπως προσπαθήσαμε να σώσουμε και το τραπεζικό κλάδο, το χρηματοπιστωτικό, ή θα αφήσουμε την αγορά να τη σκοτώσει. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να διασώσουμε αυτό το κλάδο. Τώρα για τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια μας λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατά των κρατικών ενισχύσεων, δεν θέλει κρατικές ενισχύσεις, αλλά παγιώνει τις χρονοθυρίδες και για τα χρησιμοποιητές χρονοθυρίδες την ήθα την πληρώσουν τα αεροδρόμια. Νομίζω ότι είναι κολοσσίο λάθος ε, να φέρουμε σε αντιπαράθεση τα αεροδρόμια με τις αεροπορικές εταιρείε, γιατί οι μένουν πελάτες των ΔΕ. Οπότε όταν ε, αντιμετωπίσουν δυσκολίες οι αεροπορικές εταιρείε ε, θα θυγούν άμεσα και τα αεροδρόμια. Δεν θα πρέπει μονομερώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα των αεροπορικών εταιρείων αφήνοντας κατά μέρος το πρόβλημα των αεροδρομίων. Όποια και αν είναι η λύση που θα επιλέξουμε, όποια και αν είναι, της Επιτροπής ή του Πάολο Κώστα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ε, τροποποιήσεις από τις αεροπορικές εταιρείε. Αν εμείνουμε στο 80-20, την απάντηση μας την έδωσε ο ο Στόκμαν. Θα, φυσικά θα χρησιμοποιήσουν τις καλύτερες, πιο επικερδείς χρονοθυρίδες και θα αφήσουν τις υπόλοιπες, ξεκινώντας από τις περιφερειακές. Θα διαφυλάξουν τις επικερδέστερες χρονοθυρίδες και στις περιφερειακές μεταφορές θα είναι που θα έχουμε προβλήματα. Θα κρατήσουν ε, τις πιο ενδιαφέρουσες χρονοθυρίδες και θα απαλλαγούν από τις λιγότερο προσοδοφόρες. Αν παγώσουμε το μέτρο, αν ε, αναστείλουμε την ρήτρα, την ήθε την πληρώσουν τα αεροδρόμια. Γιατί θα χρειαστεί να καταργήσουν πολλές ε, αεροπορικές ε, γραμμές οι αεροπορικές εταιρείες, γιατί δεν θα ε, θέλουν να κυκλοφορούν άδεια τα αεροπλάνα τους. Αντιλαμβάνομαι την οργή των άλλων κλάδων που λέει ότι αν, πληγεί, ε, αν πληγούν οι αερομεταφορές θα θυγούν και τα αεροδρόμια. Δεν θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε μόνο με τις αεροπορικές εταιρείε, αλλά και με αυτές και το συντομότερο δυνατό. Ας ε, μην ενδίδουμε τώρα σε αυταρέσκειες. Κι εγώ είμαι υπέρ της κοινοβουλευτικής αυταρέσκειας και του κοινοβουλευτικού εγωισμού και καλό είναι να ευλογούμε τα γένεια μας, αλλά τώρα έχουμε κρίση και είναι έκθετες οι αεροπορικές εταιρείε. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ώστε να τεθεί το μέτρο το συντομότερο δυνατό σε ισχύ για το 2009 και 2010. Και δεν πιστεύω ότι θα είναι μεταβατικό αυτό το μέτρο. Γιατί πιστεύω ότι άλλο η τελευταία κρίση και άλλο οι δύο προηγούμενες. Δεν έχουμε ούτε την 11η Σεπτεμβρίου, ούτε την κρίση του 2003. Οπότε, συνάδελφοι, θα πρέπει να συμφωνήσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, κυρίω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε πώ θα παρακολουθήσουμε αυτή την κρίση. Εγώ πιστεύω ότι καλό θα ήταν να στήσουμε μια ad hoc επιτροπή παρακολούθηση τη χρήση με Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξετάσουμε πρώτα τα στοιχεία που δεν τα έχουμε ακόμη συγκεντρώσει. Για να δούμε πώ θα διορθώσουμε τα μέτρα που έχουμε θεσπίσει γιατί η κατάσταση είναι ευμετάβλητη και για πολλούς μήνες θα μείνουμε απληροφόρητοι. Ίσως ε, υποβάλει νέα πρόταση κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα τη δει για πρώτη φορά η νέα Επιτροπή Μεταφορών το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οι περισσότεροι θα είναι καινούριοι, θα ξέρουν τι τους γίνεται. Ευτυχώς μερικοί θα συμμετέχουμε και πάλι στην Επιτροπή Μεταφορών. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παρακολούθηση εφαρμογής αυτών των μέτρων για να δούμε αν λειτουργούν αποτελεσματικά, τι παρενέργειες έχουν. Και επίσης να ζητήσουμε έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον αντίκτυπο της κρίσης στα αεροδρόμια για να διαμορφώσουμε γνώμη και για αυτό το θέμα. Και φυσικά το γοργόν και να έχει. Και θα δούμε αν δεχτούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό θα το κάνουμε υπό επιφυλάξεις. Oh. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πρέπει να παρεκτραπούμε στη συζήτηση. Γιατί η συζήτηση δεν έχει στόχο την τροποποίηση της ουσίας του κανονισμού θέλουμε να κάνουμε μια αξιολογική κρίση επί μια συγκεκριμένη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έκτακτη. Έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα, προσωρινό χαρακτήρα και υποβάλλεται εν μέσω μια αναφυσβήτητης κρίση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ναι ή όχι. Όχι επί της ουσίας. δεν είναι να τροποποιήσουμε ένα σύστημα. Υπάρχουν προηγούμενα και αναφέρθηκαν εδώ και από τον πρόεδρο ε, και έχουμε περιπτώσεις εφαρμογή τέτοιου συστήματος. Υπάρχει και μια νομική διαδικασία και αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να ληφθούν κατεπηγόντως αποφάσεις με τη συνοπτική διαδικασία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε αν υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση με τη μορφή που υποβάλλεται. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε ανεφόρον την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόνο έτσι θα είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της. Και όταν λήξει η περίοδος αυτή, τότε θα κρίνουμε αν έχει νόημα η συνέχισή της. Αλλά ήδη από τώρα θα πρέπει να δούμε θα την αποφασίσουμε ή όχι. Γιατί όλα αυτά τα ημίμετρα, όλα αυτά τα ευαλωβατικά μέτρα που προτείνουν ορισμένοι, δεν πρόκειται παρά να επιτείνουν τη σύγχυση, θα προκαλέσουν ακαδημαϊκές συζητήσεις και σίγουρα δεν θα έχουν αποτελεσματικότητα η θέση μου είναι απερίφραστα και αναφανδόν υπέρ της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι τη δυσφορία και του Προέδρου και του συντονιστή μας και με εντυπωσίασε που ο συντονιστής φαίνεται να υποστηρίζει μια ανεξέλεγκτη αγορά, ενώ στόχος μας είναι να την ε, ελέγξουμε κάπως. Σίγουρα η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου και η οικονομική κρίση είναι παγκόσμια. Ήδη ε, οι αεροπορικέ μεταφορέ και μετά την 11η Σεπτεμβρίου αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Μην ξεχνάτε ότι και την αυτοκινητοβιομηχανία τη στηρίζουμε, γιατί πρόκειται για κλάδου ε, με τεράστιο οικονομικό βάρος και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Άλλωστε δεν έχουμε εδώ αντιπαράθεση μεταξύ μεγάλων και μικρών αεροπορικών εταιριών. Μπορεί ορισμένες εταιρείες να μην έχουν συνδικαλιστικές πρακτικές αξιέπαινες, αλλά εδώ μιλούμε ουσιαστικά για όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να εμπλακούμε σε τέτοιες αντιπαλότητες. Ό,τι αφορά τα περιφερειακά αεροδρόμια, πραγματικά με σοκάρει αυτό που προτείνεται, γιατί υπάρχουν κάποιες πιο μαχητικές ε, αεροπορικές εταιρείες κατά της εξαίρεσης, αλλά τα περιφερειακά αεροδρόμια περιμένουν από τα κεντρικά αεροδρόμια μια λύση και τα κεντρικά αεροδρόμια νομίζω ότι ουσιαστικά θα τα κεντρικά αεροδρόμια θα εγκαταλείψουν τα περιφερειακά. Δεν νομίζω ότι με τη θέση αυτή προς το παρόν ε, αντιμετωπίζονται δυσμενώ τα περιφερειακά αεροδρόμια, θα πρέπει τα δικά τους προβλήματα να, τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Άλλωστε τα περιφερειακά αεροδρόμια και η στήριξή του σχετίζεται με τι κρατικέ ενισχύσει. Ενώ η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάχθηκε κατά των κρατικών ενισχύσεων. Αν θέλει να υπαναχωρήσει, πολύ ευχαρίστω. Παρόλο που, όπω είπε ο κύριο Αλμπερτίνη, έχουν άλλα προβλήματα εξαιτία τη υπερβολική τους ε, ε, επιτυχία. Είναι κατά κάποιο τρόπο θύματα τη επιτυχία τους και τη συμφόρης που αντιμετωπίζουν. Πάντως, ε, οι αεροπορικέ εταιρείε βρίσκονται στην καρδιά του αεροπορικού κλάδου και θα πρέπει εν ώψη και των εκλογών να δείξουμε στου πολίτε ότι είμαστε ικανοί να αντιδρούμε αμέσω σε μια κατεπίγουσα και έκτακτη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κύριε Σαββαρή, μπορεί να είναι παρατεταμένη η κρίση, αλλά οι κινήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των αεροπορικών εταιριών και προσπάθειες αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών μας υποχρεώνουν στο να εξετάζουμε και άλλα μέτρα. Αλλά αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γενικότερη συζήτηση για τι χρονοθυρίδε. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να το εξετάσουμε. Εδώ έχουμε μια κατεπίγουσα κατάσταση και καλούμαστε να λάβουμε πάρα αυτά μια θέση. Ευχαριστώ. Καλώς. Δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρατηρήσεις σας και τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Δεν θα ήθελα να κάνω κρίση σε περί συμπεριφοράς ε, ορισμένων, γιατί έτσι θα χαλάσουμε την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ μας και θα ήταν κρίμα τελευταία συνεδρίαση. Και νομίζω ότι έχω απογοητευτεί λίγο γιατί φαίνεται ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, αν γίνει η πρόταση καλώς, αντιμετωπίζουμε λοιπόν με τροποποίηση στα πλαίσια τη εξουσία που έχει το Κοινοβούλιο σαν συνομοθέτη. Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνει πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απομοιζόμαστε τι ευθύνε μα. Δεν λέμε ναι ή όχι, έχουμε ευθύνε, δεν κάνουμε ερμηνεία απλώ. Αυτά που αναφέρονται. Εντάξει. Πώς να το πω, πώς να το πω. Όλα αυτά που υπόθηκαν. ασχολιόμαστε με τι αεροπορικέ εταιρείε. Αύριο αλλάζουμε τι χρονοθυρίδε, μετά αλλάζουμε τα τέλη αεροδρομίων κλπ. Όλα αυτά είναι αναλυτικό σφάλμα. Το αναλυτικό σφάλμα μπορούμε να κάνουμε τώρα. Η κρίση είναι διαφορετική. Είναι η κρίση όλων, όχι μερικών. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τομεακά. Δεν είναι ένα πρόβλημα ενό μικρού τομέα. Είναι τουλάχιστον όρου του τομέα των αερομεταφορών που αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα. Πρέπει να έχουμε τη βούληση να είμαστε φάνταστοι, να έχουμε τη δύναμη, το θάρρος, μπορώ να το πω και αυτό, να έχουμε το θάρρος, να αντισταθούμε σε κάποιες αλαζονικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται αυτές τις εβδομάδες, που ξεπερνούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Ποτέ δεν έχουμε επηρεάσει, αλλάξει τόσο σημαντικά συμφέροντα. Κύριε Στόκμαν, το πρόβλημα το δημιουργήσαμε εμείς δεχθήκαμε έστω και παθητικά ένα δημόσιο αγαθό, οι χρονοθυρίδες να γίνουν αγαθό ιδιωτικό. Δεχθήκαμε εμείς, οι θεσμοί, τα θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την που δίνει, το δεχθήκαμε. Η ζημιά από εκεί ξεκινάει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το πρόβλημα, δεν το έλυσε. Μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτήν τη στιγμή να λύσουμε το πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό το κλίμα. Εγώ, αν ίσχυε αυτό με δύο γραμμέ που θα έγραφε ο κύριο Στόκμαν, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τον κανονισμό όσον αφορά τι χρονοθυρίδε τώρα. Και τώρα είναι η στιγμή να γίνει. Αυτή τη στιγμή ο κόσμο αισθάνεται ότι χρειάζεται να αλλάξει κάτι τι. Να μιλήσουμε αργότερα πότε. Δεν θα μιλήσουμε ποτέ αν δεν μιλήσουμε τώρα. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή είναι μια μάχη που πώς να το πω που δεν μου επιτρέπω να διανοηθώ καν ότι θα την πολεμήσω τη μάχη αυτή μόνος μου αλλά είναι και θέμα υπερηφάνειας του Κοινοβουλίου. Εγώ έτσι αλλιώς το βλέπω αυτό. Δεν είναι πρόβλημα να πούμε ναι ή όχι. Έχουμε προτάσεις πάρα πολλές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν έχουμε δεχτεί σε δύο λεπτά. Αλλά νομίζω ότι είναι άδικη. Λοιπόν, θα υπομιστούμε τις ευθύνες μας, ναι ή όχι και χωρίς να χρονοτριβούμε μέσω της διαδικασίας. Διότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 22 ψηφοφορίες στην Επιτροπή. Είναι προφανές ότι δεν θα έχουμε ομοφωνία επί αυτών που θα προτείνω, άρα 22 θα το ψηφίσουμε το θέμα στην Επιτροπή και μετά θα γίνουν συνδιαλλαγές με το Συμβούλιο. Να μην χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο λοιπόν, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε για 20 μέρες ανοιχτή τη συζήτηση. Μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάσουμε κάποιε ιδέε, να κάνουμε κάποιες προτάσεις για να αλλάξουμε λίγο αυτή την κατάσταση. Ναι, Ιού, ή πρέπει να φοβόμαστε να τρομοκατηθούμε και να πούμε ότι δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα υπάρχει. Μέχρι χτε ο κύριο Γιαζεμπόφσκι θεωρούσε ότι ήταν λογική η πρόταση. Εντάξει, άμα θεωρεί ήταν λογική πια, τι να κάνουμε. Δεν έχω εφεύρει εγώ την ε, ε, πρόταση αυτή. Εγώ συζήτησα, την οικοδόμησα. Ξαφνικά δεν ισχύει πια. Ο καθένα από εμά έχει το δικαίωμα ε, να βλέπει οράματα, όπω καθοδόν προ τη Δαμασκό, ο Παύλος, ο Πόστο Παύλος Εντάξει, όταν βλέπουμε οράματα και αλλάζουμε γνώμη, εντάξει. Όμω, τι να πω. Να το πω έτσι τώρα, κλείνοντα. Έλεγα ο παππού μου, που ήταν και χωρικό, ότι όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις και θα νικήσει όχι, καλό είναι να κάνεις το δίκιο. Ε, λοιπόν, τέλος της συζητήσεως, εγώ θα κάνω τι θεωρώ δίκαιο και σωστό. Πέρα στις συζητήσεις.